Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυρίσω την έναρξη της πρώτης μας συνεδρίασης ε, το 2017. Με μικρή καθυστέρηση ξεκινάμε. Αλλά έπρεπε να σας δώσω λίγο χρόνο να ανταλλάξετε ευχές. Και θα ήθελα και εγώ να σας ευχηθώ ευτυχισμένο το νέο έτος, το 2017. Να πάνε όλα καλά. Και να ξεκινήσουμε από τα διαδικαστικά, πριν καλωσορίσω τους καλεσμένους μας. Καταρχήν έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Δεν βλέπω παρατηρήσεις, οπότε την εγκρίνουμε. Έχουμε και αναμετάδοση απευθεία από το διαδίκτυο τη συνεδρίασης και διερμηνία σε 20 γλώσσε. Με εξαίρεση τα εσθονικά, μαλτέζικα, σλοβακικά και γοεδελικά. Α εγκρίνουμε και τα πρακτικά της συνεδρια 26 26-29 Σεπτεμβρίου 2016. Ακολουθούμε την γνωστή διαδικασία και περνάμε στο κυρίως θέμα της ε, απογευματινής ημερήσιας διάταξης την ακρόαση με θέμα τα συμπεράσματα της ειδικής ομάδας εργασίας για τις ε, αγορές των γεωργικών προϊόντων. Κυρίσω την έναρξη αυτής της ακρόασης, καλωσορίζοντας ε, θερμότατα τους καλεσμένους μας, τους εμπειρογνώμονες και τους ευχαριστώ ταυτόχρονα για την αποδοχή της πρόσκλησης και για την παρουσία τους. Ε, ξεκινώ από τον Επίτροπο Χόγκαν που ήταν και πρωτεργάτης ε, αυτής της ε, προσπάθειας και της σύστασης αυτής της ειδικής ομάδας εργασίας. Επίσης, να καλωσορίσω τους εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους εκπροσώπους ε, του Συμβουλίου, της ΚΟΠΑ ΚΟΖΕΚΑ και όλους τους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων. Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σε αυτή την πολύ σημαντική δημόσια ακρόαση. Καλωσορίζω και τους ευρωβουλευτές, τους συνεργάτες τους, τους βοηθούς τους. Και περνάμε στο θέμα τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Αγροεπιστηστικού Κλάδου στις παγκόσμιες αγορές. Μια συμμετοχή που δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες και δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα τον καθιστά πιο ευάλωτο στους εξωτερικούς παράγοντες και στα προβλήματα κυρίως της αστάθειας ε, των ε, συνθήκων των παγκόσμιων αγορών και κυρίως τις διακοιμάσεις, τις απότομες διακοιμάσεις των τιμών των γεωργικών προϊόντων. Το έχουμε δει αυτό και σε εκθέσεις της Επιτροπής μας. Οπότε ε, έχουμε μια εξωτερική κατάσταση και εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη, τα γεωρικά μας προϊόντα, αλλά έχουμε και εσωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αγροεπιστηστική μας ε, βιομηχανία. Έχουμε και εσωτερικά προβλήματα που επηρεάζουν τις αγορές των γεωρικών προϊόντων. Οπότε εδώ ε, θα εξετάσουμε διάφορα θέματα όπως τη διαφάνεια της αγοράς, την πρόσβαση των γεωργών στα χρηματοπιστωτικά μέσα και στην χρηματοδότηση, στις αγορές των ε, συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης, Futures Markets και θα δούμε τις διάφορες σχέσεις μεταξύ των κρίκων της, της τροφικής ε, απιστιστικής αλυσίδας. Και προτείνουμε και κάποιες ε, νομοθετικές ρυθμίσεις. Όλα αυτά τα θέματα ήταν το αντικείμενο της ομάδας εργασίας αυτής για τις αγορές γεωργικών προϊόντων. Η ομάδα αυτή εργασίας, η ειδική ομάδα εργασίας, απαρτίζεται από 12 μέλη, από πεπειραμένους εμπειρογνώμονες ε, και έγκριτους ε, καλεσμένους, έγκριτους ε, ειδικού της διατροφικής αλυσίδας. Χθες δυστυχώς ενημερωθήκαμε ότι ο κύριος Βέρμαν δεν θα μπορέσει να λάβει μέρος στη συνεδρίασή μας. Τον αντικαθιστά όμως ο κύριος ε, Χέλφριτ Γκίζεν, που ήταν ε, πρώην εκτελεστικός διευθυντής ε, του Συμβουλίου της, του Συνεταιρισμού Κρέατος Westflies. Επίσης έχουμε και την κυρία Νίκο Γιούχας, επίσης εκτελεστική διευθύντρια. Και ο κύριος Γκίσεν θα κρίνει ε, αν θα δώσει το λόγο και σε άλλα μέλη της ειδικής αυτής ομάδας εργασίας, αν το κρίνει απαραίτητο. Όπως σας είπα, ο Επίτροπος Χόγκαν ενθάρρυνε την Επιτροπή μας να συμβάλλει με τις παρατηρήσεις της στο έργο αυτής της ε, ειδικής ομάδας εργασίας, αυτής της Task Force και μάλιστα με τις διάφορες εκθέσεις μας ε, παρακολουθούμε τις εργασίες αυτής της Task Force ε, εδώ και πολύ καιρό, από την έναρξη της κοινοβουλευτικής μας θητείας. Ε, αυτή η Task Force ε, παρουσίασε την οριστική της τελική της έκθεση τον περασμένο Νοέμβριο με συγκεκριμένες συστάσεις πολιτικής και συστάσεις για νομοθετικές πρωτοβουλίες. Οπότε Μία ακρόση έγινε και τη ειδική αυτή ομάδα εργασία στο Συμβούλιο Υπουργών, οπότε έχετε ήδη αποκομίσει κάποιε πρώτε εντυπώσει από το έργο αυτή τη Επιτροπή. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον Επίτροπο για να ε, μα ενημερώσει. Ευχαριστώ επί τη ευκαιρία και του διερμηνεί και το προσωπικό και σα δίνω το λόγο, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ που με καλωσορίσατε και τις ευχές για το νέο έτος, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, ενδιαφερόμενοι εκεί, εκπρόσωποι τους, κύριε και κύριοι, καταρχάς να ευχαριστήσω επιστήμως ε, τα μέλη της ομάδας Task Force για τα αγροτροφομικά, για τις εργασίες του 2016. Σίγουρα θα πιστεύετε κι εσείς ότι έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά και είναι στέρη βάση αυτή για εργασία του επόμενου έτους και των επόμενων ετών και ευχαριστώντα τα μέλη της Task Force θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι πολύ ασύνηθες στα θεσμικά όργανα να έχουμε εργασίες που ξεκινούν στις αρχές του έτους και που ολοκληρώνται πριν να ολοκληρωθεί και το έτος. Δεν συμβαίνει αυτό συνήθως. Χαίρομαι ιδιαίτερα που πετέυθεί αυτό. Πριν λοιπόν μπω σε λεπτομέρειες όσον αφορά την έκθεση, θέλω να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα και ελπίζω ότι μετά από κάποια δύσκολα χρόνια που περάσαμε το 2017 θα είναι καλύτερο έτος για τους γεωργούς. Βελτιώνεται η όλη κατάσταση στην αγορά και αυξάνονται οι τιμές με αργό σταθερό ρυθμό. Είδαμε τα στοιχεία για τις τιμές του νευρίου για το γάλα και αυτά μας δίνουν λόγους αισιοδοξία. Όμως θα πρέπει να επαγρυπνούμε όσον αφορά την αγορά των τροφίμων για το 2017 διότι η ανάκαμψη είναι εύθραυστη Ελπίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι σημαντικό έτος για τις γεωργικές πολιτικές το 2017 και προσβλέπω συνεργασία μαζί σας για να συνεχίσουμε να πλουστεύουμε την ΚΑΠ, να γίνει πιο αποτελεσματική η ΚΑΠ και να ταιριάζει στις ανάγκες των γεωργών μας. Μπορώ να βασιστώ στην επικοδομητική προσέγγιση τη Επιτροπή σα, πιστεύω, σε αυτή την προσπάθεια, ώστε τελικά η πολιτική μα να πετυχαίνει του βασικού στόχου προ όφελο των αγροτών μα. Βλέποντα την έκθεση που έχουμε μπροστά μα, ε, την έκθεση τη ομάδα Κρούσο, ε, πιστεύω ότι είναι σωστό να γίνεται αυτή η συζήτηση στι αρχέ του έτου. Δυστυχώ, όπω είπε και ο Πρόεδρο, ο κ. Βίρμαν δυστυχώ δεν δύναται να είναι εδώ λόγω γρήπη. Δεν έχει κάτι πιο σοβαρό, αλλά θα βελτιωθεί η κατάστασή του. Με τα χαρά λέγω ότι η Health Edition είναι εδώ για να εκπροσωπήσει την ομάδα κρούση και βεβαίω έχει και τη βοήθεια και των μελών τη ομάδα κρούση που είναι εδώ. Οι έξι εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα ήταν πάρα πολύ δραστήρια τις εβδομάδες και θέλω να διατηρήσουμε αυτή την ένταση των εργασιών του 2017. Είναι ένας άλλος σταθμός τώρα στην προσπάθεια βελτίωσης της θέσης του Γεωργού στον αγροτροφημικό τομέα. Τον Νοέμβριο λοιπόν η Task Force παρουσίασε τα πορίσματά της και ήταν πάρα πολύ σημαντικό βήμα αυτό εγκαίρως υπέβαλα την έκθεση, δώσανε πάρα πολλές λεπτομέρειες, εύληπτες. Είναι πρακτική η έκθεση αυτή. Η ανεξαρτησία της τεχνογνωσίας της Task Force δίνει μεγάλη εξοπιστία στο όλο έργο. Και είχαμε θετικές δραστηρι... ε, αντιδράσεις τις και αυτό δείχνει πόσο ποιοτική είναι η έκθεση. Το 2015 και το 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε τους γεωργούς της του υποστήριξε όσον αφορά τι δυσκολίε που δημιούργησε η αγορά και απειλούσε τη βιωσιμότητά του. Τα θεσμικά όργανα υιοθέτησαν τρία πακέτα αλληλεγγύη, 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ συμπληρωματικά η βοήθεια και 22 μέτρα. Και έτσι δείξαμε ότι είμαστε πρόθυμοι, βραχυπρόθυμοι να κινηθούμε και μέσω εξαιρετικών μέτρων, εκτάκτων μέτρων, λόγω σοβαρών δυσκολιών τη αγορά. Θέλω λοιπόν να παραδεχτώ το ότι μα στήριξε το Κοινοβούλιο, στήριξε του γεωργού τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω στο Κοινοβούλιο, ήταν επικοδομητική υποστήριξη στι προσπάθειε επίση Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά κυρίω με τι κατεξοδότητε συμπράξει, εφαρμοστικέ πράξει και όλε τι συζητήσει για το πακέτο και τα πακέτα αλληλεγγύη. Όμω η συνεχή υποστήριξη μέσω πακέτων σε αυτή την κλίμακα και σε τέτοια έκταση δεν είναι κάτι βιώσιμο στο μέλλον, κυρίως υπό το φως των άλλων πολιτικών και δημοσιονομικών προβλημάτων που γνωρίζεται και αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, μαζί με αυτά τα πακέτα, που όπως ανέφερα ανέρχονται στα 2,5 δις ευρώ για να υποστηρίξουμε τους ε, γεωργούς μας, θα βρούμε νέους τρόπους για βελτιώσεις διαθροτικές για να αποφύγουμε την επιβολή εκτάκτων μέτρων στο μέλλον, όπω όλοι θα συμφωνείτε, υπάρχει κατ' ανάγκη να βελτιωθεί η αντοχή του γεωργικού μα τομέα και θεωρώ ότι αυτό είναι μια από τι μου στα πλαίσια τη ανακοινώσεώ μου για το 2017. Ο κ. Γκίσεν θα σα δώσει λεπτομερή επισκόπηση των συστάσεων τη ομάδα Κρούς αργότερα. Ουσιαστικά λοιπόν οι συστάσει καταλήγουν στο πόρισμα ότι το πλαίσιο πολιτική για την υποστήριξη θα πρέπει να βελτιωθεί όσον αφορά τον εφοδιασμό σε τρόφιμα και καλή έκθεση για νέου κανόνε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να καλυφθούν κάποιε αθέμητε πρακτικέ στο εμπόριο, καθώ και την ε, εφαρμογή αποτελεσματικών καθεστώτων επιβολή των μέτρων στα κράτη-μέλη μέσω τη χρήση ενό διαμεσολαβητού που θα κρίνει, ενό κριτή. Ε, χρειάζεται αύξηση τη διαφάνεια αγορά. Θα πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των γεωργών. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση των γεωργών στη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να βελτιωθεί ε, η χρήση εργαλείων αντιμετωπίσεω των κινδύνων. Σε σχέση με τι αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ, η έκθεση συστήνει ότι νομοθεσία πλαίσιο θα πρέπει να θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να καλυφθούν κάποιε βασικέ πρακτικέ αθέμητε, όπω μέγιστε με περίοδοι πληρωμή και θα πρέπει να υπάρχουν καθεστώτα σωστά εφαρμογή των μέτρων σε κάτι μέλη και να υπάρχει κάποιο αρμόδιο φορέα γι' αυτό. Τα ευρωβουλευτέ ηγήθηκαν στην προσπάθεια ήδη που κατεβλήθη με συστάσει ένθερμε προ σωστή κατεύθυνση. Και η έκθεση υιοθετήθηκε πέρσι τον Ιούνιο με μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβούλιο... 600 ψήφοι με 38 ήταν η ψηφοφορία και ζητήθηκε να αναλυθεί η νομοθετική πρακτική, να αποτελεμηθεί η αθέμητη πρακτική όσον αφορά την σε τρόφιμα. Και το Δεκέμβριο του 2016 η Ποσλοβακική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ομόφωνα συνεπέρανε το Συμβούλιο ότι πρέπει να ισχυθεί η θέση των γεωργών στην τροφιμική αλυσίδα ζητώντας να γίνει αξιολόγηση συνεπιών ε, το ταχύτερο δυνατόν στα πλαίσια νομοθεσίας πλαισίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως ούτως ώστε να κρυθούν παρανόμες κάποιες αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Οι υπουργοί επίση προσυπόγραψαν, αν θέλετε, το θέμα αυτό για μεγαλύτερη διαφάνεια και στα περιθώρια των τιμών και μεγαλύτερη διευκρίνηση των ε, ορισμών για να υπάρχει καλύτερη συνεργασία σε επίπεδο παραγωγών και να είναι δίκαιη αντιμετώπιση των γεωργών όσον αφορά τα προϊόντα του, τι τιμέ για τα προϊόντα του. Το Δεκέμβριο του 2015 και του 2016, εκπρόσωποι τη αγροτοφημική αλυσίδα και όλα τα, από όλα τα κάτι μέσα Ευρωπαϊκή Ενώσεω πήγαν στο φόρουμ ψηλοπιπέδου για την καλύτερη λειτουργία τη ε, αλυσίδα ε, αφοδιασμού και ήμουνα και εγώ παρόν και εκεί η μεγάλη πλειοψηφία των εμπλεκομένων φορέων, κυρίω ε, το τομέα μεταπίση των τροφίμων, εξέφρασαν την υποστήριξή του ότι θα έπρεπε να υπάρξει νομοθεσία πλαίσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θεωρίζει ελάχιστε προδιαγραφέ για τι αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ. Ο Επίτροπο Μπιενκόλσκα έδωσε σαφέ μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεσμευμένη να αντιμετωπίσει του φραγμού τη ενιαία αγορά για τα τρόφιμα. Ετώνησε ότι δεν θα υπάρχει θέση για θέμητε εμπορικέ πρακτικέ σε μια σύγχρονη αλυσίδα εφοδιασμού σε τρόφιμα. Κυρίε και κύριοι, λοιπόν, όλα αυτά τα μηνύματα δείχνουν τη σωστή κατεύθυνση και τώρα από εμά εξαρτάται που διαμορφώνουμε την πολιτική να ακολουθήσουμε τα επόμενα βήματα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε συνετά και προσεκτικά. Δεν υπάρχει ένα μέτρο το οποίο θα είναι πανάκια για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων. Υπάρχουν σαφεί δρόμοι που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να καταλήξουμε σε καλύτερο μέρο. Συνεχή συντονισμένη δράση απαιτείται. Έτσι μπορούμε να έχουμε πιο ανθεκτική γεωργία και πιο αποτελεσματική και υγιεινή δυνατότητα χωρισμού σε τρόφιμα. Η Task Force θεωρεί ότι έχει στρατηγική σημασία η δικαιοσύνη στον τομέα παραγωγή τροφίμων για να επιβιώσει η ύπεθρο, γιατί είναι ο ζωντανό ιστό τη υπαίθρου η Γεωργία. Αυτό πιστεύω ότι το πιστεύετε και εσεί εδώ στην ε, Επιτροπή Γεωργία και χαίρομαι που η Επιτροπή σα και κύριε και ε, Πρόεδρε διοργανώσατε αυτή την ε, συνάντηση εδώ. Καλέσατε τον κύριο Κίσα να παρουσιάσει συμπεράσματα τη Task Force και Καλέσατε και ένα πάνελ ειδικών και έτσι έχουμε το ιδεώδες βήμα για να συζητήσουμε το θέμα. Να δούμε πώς θα μεταφραστεί το έργο της Task Force από προτάσεις να μεταμορφωθεί σε πραγματικότητα. Προσβλέπω λοιπόν στις συζητήσεις και θα έχουμε τη δυνατότητα μαζί με τον, Κίσεν, τον κύριο Γκίσεν να δώσουμε και απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις που θα ακολουθήσουν την παρουσίαση των θεμάτων. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, πριν περάσουμε στην ακρόαση των εμπειρογνωμόνων μας, θα ήθελα να καλωσορίσω και τους ε, δημοσιογράφους που είναι παρόντες ε, μετά από πρόσκληση της ε, κυρίας Κέστιγκερ. Η κυρία Κέστιγκερ είναι πολύ δραστήρια ευρωβουλευτής με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και θα συγκεντρώσουμε για αυτήν την ακρόση πλούσιο υλικό Περνάμε τώρα στην ακρόαση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκίσεν για να μας παρουσιάσει την έκθεση της ε, Ειδικής Επιτροπής, της Ειδικής Ομάδας Εργασίας, της Task Force. Μετά θα ακούσουμε τον κύριο Μάρτιν Μέριλτ, τον πρόεδρο της ΚΟΠΑ, κατόπιν τον κύριο Γιώζεφ Πλάνκ, που είναι γενικός ε, γραμματέας της, του Αυστριακού Γεωργικού Επιμελητηρίου, κατόπιν τον κύριο Μέριχ Ρέιμοντ, που είναι πρόεδρος της ε, Βρετανικής Ένωσης Γεωργών, ε, και μετά στον κύριο Γιώστ Πένιγκς, που είναι καθηγητής οικονομικών και μάρκετινγκ στα πανεπιστήμια του Μάστρεκ και του Βάγενιγκεν. Θα δώσω πρώτο το λόγο στον πρόεδρο Γκίσεν για να μας κάνει την παρουσία της, της έκθεσης της Task Force. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Κυρίε και κύριοι, καλή χρονιά για από μένα. Και βεβαίω μια καλή παρουσίαση ξεκινάει με μια ωραία εικόνα, κάτι το οποίο νομίζω έχετε ήδη μπροστά σας, τον Επίτροπο με τους εμπειρογνώμονες της ε, Task Force. Είχαμε λοιπόν πέρσι στις 13 Ιανουαρίου μια σχετική συνεδρίαση και είχαμε την πλήρη υποστήριξη Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και νομίζω πως είχαμε ένα επιτυχημένο μείγμα των ειδικών ε, από διάφορους κλάδους της επιστήμης, ε, της διοίκησης, των κρατών μελών, ε, των διαφορών κλάδων ε, της ε, διατροφικής βιομηχανίας. Νομίζω ένα επιτυχημένο μείγμα, ε, καθώς βεβαίως και ένα πάρα πολύ καλό συντονιστή, τον κύριο Φέρμαν, καθώς χωρίς αυτόν δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα των 70 σελίδων. Θα ήθελα να το χειθώ επί τη ευκαιρία και καλή ανάρρωση. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στο πλαίσιο των ε, όσων ε, κάναμε. Κάποια από τα πράγματα αυτά ήδη αναφέρθηκαν. Είχαμε το Συμβούλιο του 2015, το Συμβουλίο Γεωργίας, το οποίο αναφέρθηκε και στην κρίση του γάλακτος ε, και βεβαίως στόχος ήταν να δούμε την κατάσταση σε διαφορούς κλάδους και υπήρχε και η ομάδα εργασίας ειδικών υψηλού επίπεδου και κατέστη σαφές ότι θα έπρεπε να δούμε τις αγορές, την, την αλυσίδα δημιουργίας ε, αξίας για να δούμε πού και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε, να ενισχύσουμε την θέση των αγροτών και τον ρόλο των αγροτών στις αγορές. Και πράγματι θεωρούμε ότι εδώ πέρα απαιτείται κάποια δράση και είχαμε 8 συνεδριάσεις ε, και με την ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου και το αποτέλεσμα βεβαίω ήταν η τελευταία συνεδρίαση στις 3 Νοεμβρίου και η παρουσίαση της έκθεσης στις 14 Νοεμβρίου του 2016, έκθεση η οποία βεβαίως απευθύνεται σε όσο δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό χρηστών. Προσπαθήσαμε να κάνουμε συγκεκριμένες ε, συστάσεις χωρίς βεβαίως να περιλάβουμε τα πάντα σε αυτό το κείμενο. Αυτό λοιπόν είναι το έγγραφο το οποίο έχετε μπροστά σας και ελπίζω να μπορέσετε να το διαβάσετε. Νομίζω ότι είχαμε ήδη μια πρώτη θετική αντίδραση. Να περάσω στο επόμενο σημείο, η σύλληψη, η γενικότερη συζήτηση κινήθηκε στο πλαίσιο του ότι η ε, μεταρρύθμιση αυτής της κοινή γεωργικής πολιτικής είναι η βάση της ε, πολιτικής μας. Έχουμε το θέμα ακριβώς της αποσύνδεσης ε, από την παραγωγή, να δώσουμε δηλαδή περισσότερο ρόλο στις αγορές. Αν δείτε παραδείγματος χάρη το τι γίνεται με το γάλα, το αποκτηρωμένο και το βούτυρο. Νομίζω πως έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα στο πακέτο των μέτρων. Όχι μόνο για αυτό τον λόγο, αλλά παράλληλα με αυτό θα έλεγα οι αγορές έπαιξαν τον ρόλο τους, αλλά νομίζω πως κατά τη του περασμένου έτους ε, είδαμε τον ρόλο τους. Ο ρόλος των αγροτών εδώ πέρα. προσπαθούμε ακριβώς να δούμε ποια θα είναι η μορφή της οργάνωσης που θα έχουν ως συνεταιρισμοί, ως ε, ενώσεις παραγωγών να αποκτήσουν μεγαλύτερο βάρος σε αυτή την αλυσίδα και ε, παρόλα αυτά ήταν σαφές ε, πως η κατάσταση αλλάζει, έχουμε την, τις νέες πτυχές της κλιματικής αλλαγής. Τα τελευταία χρόνια είχαμε σημαντικές διαφορές ε, στις σοδιές στη Ισπανία, στη Γαλλία και βεβαίω πρέπει να δούμε και τη διαχείριση του περιβάλλοντος κάτι το οποίο βεβαίω αποτελεί και ένα νέο, μια νέα κινητήρια δύναμη όσον αφορά την επανεξέταση του ρόλου των αγροτών των οποίων είπαμε ότι θέλουμε να ενισχύσουμε να γίνει η θέση τους πιο αισθητή. Γι' αυτό εστιάσαμε σε 7 ε, κλάδους. Ο πρώτο ήταν ε, το ότι στείλαμε ένα μήνυμα με την διαφάνεια της αγοράς, με τη διαχείριση κινδύνου, με τις προθεσμιακές αγορές ε, και βεβαίως το θέμα των συμβάσεων που θα πρέπει να και αποκτούν όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία είναι πλέον γραπτές συμβάσεις δεσμευτικές, έχουμε βεβαίως και τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, ε, κάτι το οποίο οπωσδήποτε δεν αφορά μόνο τον ε, τομέα των ε, τροφίμων, απλά τον αφορά στο μέτρο στον οποίο είναι επιχειρηματική δραστηριότητα και βεβαίως έχουμε και το θέμα των συγκρούσεων και μεταξύ ακόμα των γενικών διευθύνσεων, π.χ. της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και τη γενικότερα του δικαίου του ανταγωνισμού. Ναι, δηλαδή το να καθορίζουν οι αγρότες τις τιμές ε, είναι και αυτό ένα ζήτημα και είναι κάτι το οποίο ε, γίνεται βεβαίως ε, ανεκτό Και βεβαίω ε, τίθεται και το τελευταίο ζήτημα, η πρόσβαση στην χρηματοδότηση, κάτι το οποίο εξαρτάται και από το επίπεδο της ρευστότητας και των επιτοκίων. Τώρα για να μπει μια τάξη στις ιδέες που έχουμε σε αυτές τις 70 σελίδες θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα σημείο στο οποίο προτείνουμε ρύθμιση. Μια απόφαση, απόφαση για τα σημεία που βλέπετε εδώ πέρα με κόκκινο στο 1, στο 5 και στο 6. Στο 1 βλέπουμε κάποια πρόοδο, βλέπουμε πως τα καλύτερα στατιστικά στοιχεία στον τομέα του, υπάρχουν στον τομέα του γάλακτος ε, και στον τομέα του κρέατος και θα πρέπει να έχουμε έγκυρα στατιστικά στοιχεία και αλλού, σε άλλους κλάδους. Βλέπουμε παραδείγματο χάρη το Αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας τι δεδομένα και τι ποιότητας δεδομένα έχει. Είναι πάρα πολύ πολύτιμα αυτά τα στοιχεία. Ακριβώς αυτός ο κλάδος θα πρέπει να αυξήσει την διαφάνεια της αγοράς και αυτό έχει σημασία και για τον μεμονωμένο αγρότη. Όταν έχει πληροφορίες μπορεί να αντιδρά, μπορεί να κινηθεί ανάλογα με τις αγορές. Επίσης πάμε στο 5 οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές, το ανέφερε ήδη ο Επίτροπος, είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Η πρόταση είναι να ρυθμίσουμε στο δυνατόν λιγότερο, δηλαδή να θέσουμε ένα πλαίσιο, στην, ε, πλαίσιο ε, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να γίνει σεβαστός ο φόβος ο οποίος υπάρχει πολλών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ότι αν δεν δηλώσουν κάτι θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει επίσης ε, και ένας συνήγορος εδώ πέρα ο οποίος προτείνεται για ε, να ξεκινήσουμε. Βεβαίως ε, καλό είναι να ξεκινήσουμε στην αρχή με ένα καθεστώς το οποίο θα είναι εθελοντικό, αλλά εάν δεν προχωρήσει θεωρούμε πως θα πρέπει να υπάρξει κάποια υποχρεωτική ρύθμιση. Τρίτον, είμαστε στο θέμα του δικαίου του ανταγωνισμού. Να επιτρέψουμε σε αναγνωρισμένες ενώσεις παραγωγών να αποφασίζουν και να ορίζουν τιμές και ποσότητες, αλλά όχι την ποιότητα. Κάτι το οποίο συμβαίνει ήδη, παραδείγματο χάρη στην Ισπανία με το ελαιόλαδο, οι ενώσεις ε, των ε, παραγωγών θέλουν να αποθηκεύουν επί σειρά ετών ε, το ελαιόλαδο. Θεωρώ πως εδώ πέρα πρέπει να δράσουμε για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. το, το αν θα υπάρξει κάποια κοινή αποθήκευση ή κάποια κοινοτική πρωτοβουλία θεωρούν πως θα πρέπει η Κομισιόν να αναλάβει δράση. Περνάμε στο επόμενο θέμα, στην επόμενη κατηγορία θεμάτων όπου λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια διευκόλυνση να γίνουν τα πράγματα πιο εύκολα. Αυτό αφορά τα σημεία 2, το διαχείριση κινδύνου, το 3, τα προθεσμιακά συμβολία και το 4, την χρήση των συμβάσεων. Για τη διαχείριση του κινδύνου βεβαίως έχουμε τις ασφάλειες οι οποίες αφορούν ε, το χαλάζι, αφορούν ε, τις επιζωοτίες. Αυτά τα πράγματα υπάρχουν οπωσδήποτε και σήμερα. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ακριβώς ότι όλα αυτά είναι ένας ρόλος του αγρότη που είναι ένας ρόλος διαχείρισης κινδύνου. Για να πρέπει να υπάρχει όντω αυτή η ασφάλεια και βεβαίως ε, θα πρέπει να στηρίξουμε νομίζουμε και τις εταιρείες αντασφάλισης να εμπλακούν σε αυτόν τον τομέα, ειδικά όταν θα έχουμε ή στο μέλλον περισσότερα προβλήματα με τις σοδιές, όπως είδαμε και τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής, έχουμε πλέον ορατά ζητήματα και βεβαίως αυτό επηρεάζει εμέσως και τα συμβόλαια μελλοντική ε, εκπλήρωσης ε, στα οποία μπορούμε μόνο να βοηθήσουμε να μπουν περισσότερο στην αγορά. Χρειάζεται η εμπειρία των χρηματιστηρίων όπου υπάρχει ήδη ο καθορισμός των τιμάτων των δημητριακών, καθορισμός των τιμών των δημητριακών όπου οι μεγάλοι έμποροι και οι μεγάλοι συνεταιρισμοί συνεννοούνται στα χρηματιστήρια και συνάπτουν συμφωνίες μελλοντικής εκπλήρωσης. Ε, βεβαίως απέχουμε πολύ από κάτι τέτοιο στις αγορές κρέατος και γάλακτος. Βεβαίως δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τον μεσίτη εδώ πέρα στις αγορές αυτές. Έχουμε μια πολύ μικρή εμπειρία και δεν μπορούμε ακόμα να περιμένουμε θαύματα. Το επόμενο θέμα αφορά τις συμβάσεις και βεβαίως πράγματι μπορεί κάποιος ο οποίος παράγει ζαχαρότευτλα ή ένα σφαγείο ή ο κτηνοτρόφος αν θέλει να έχει ένα κείμενο δεσμευτικό για την επιχείρησή του θα πρέπει να μπορεί να το κάνει. Θα πρέπει όμως να υπάρχει ελάχιστη δυνατή ρύθμιση και ε, μην ξεχνάμε ότι στον τομέα των συνεταιρισμών πολλά πράγματα λύνονται στο επίπεδο του μέλους του συνεταιρισμού, αλλά θα πρέπει, νομίζω ότι θα πρέπει στο μέλλον οι συμβάσεις να βελτιώσουν και να σιγουρέψουν την θέση των αγροτών στην αγορά. Γι' αυτό ακριβώς ε, αξίζει το ρόλο να δούμε πώς μπορούμε να εμβαθύνουμε τον ρόλο των συμβάσεων, ποιες είναι οι πιθανές αμφιβολίες. Βεβαίως στην Ευρώπη είναι τελείως διαφορετική, ειδικά στη Δυτική Ευρώπη, διαφορετική η παράδοση με τους συνεταιρισμούς σε Γαλλία, Γερμανία, Μπενελούξ ε, σε σχέση με την Ανατολική Ευρώπη. Και βεβαίως έχουμε το σημείο 7, την πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Έχουμε φτάσει σε μηδενικά επιτόκια, οπότε είναι πολύ περιορισμένη κατάσταση σε πολλές ε, χώρες. Αλλά βλέπουμε πώς, πόσο μεγάλη μπορεί να είναι εδώ πέρα η δύναμη του προγράμματος Juncker και στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη για να ε, ενισχύσουμε ακριβώς αυτές τις πτυχές που θα πρέπει τέλος να δούμε τα πράγματα περισσότερο. Βεβαίως δεν είναι έτοιμες αυτές οι απαντήσεις ε, που σας δίνω. Είναι περισσότερο κάποια ερεθίσματα για μια συζήτηση. Που, ε, ποιο ακριβώς είναι λοιπόν το όριο της διαχείρισης κινδύνου που επιτρέπεται το κράτος να βοηθήσει μια επιχείρηση γιατί ε, είναι μια επιχείρηση ε, η αγροτική εκμετάλλευση, παραδείγματο χάρη, ναι, μπορεί να τον βοηθήσει στην κατάρτιση ε, χωρίς βεβαίως να ξεπεράσει το εμπόριο, το, το όριο αυτό το οποίο θεωρείται κρατική ενίσχυση. Το σημείο 4, Παραδείγματο χάρη, είναι η χρήση των συμβάσεων. Δεν θέλουμε όμως ε, να οδηγηθούμε σε περαιτέρω γραφειοκρατικοποίηση. Θέλουμε απλά να ενισχύσουμε τους παραγωγούς και να έχουν στα χέρια τους ένα ξεκάθαρο κείμενο το οποίο θα αναφέρει τιμή, ποιότητα, χρόνο της παράδοσης και τι γίνεται με τα γεγονότα που είναι εκτός του ελέγχου του. Αυτά. Λοιπόν και περνάμε βεβαίως και στην πρόσβαση στην ε, χρηματοδότηση. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα, αν μου επιτρέπετε να πω δύο-τρία λόγια για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Υπάρχουν αθέμητες εμπορικές πρακτικές σε όλους τους κλάδους. Και βεβαίω στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων. Εμεί δεν θέλουμε τώρα να πούμε ποιος είναι ο κακός εδώ πέρα, ούτε να μείνει κάποιος με το μουτζούρι. Αυτό το οποίο θέμε είναι να μην πληρώνονται οι αγρότες μετά από 60, 70, 80 μέρες. Όταν μιλάμε για φρέσκα προϊόντα θα πρέπει να γίνονται και γρήγορα οι πληρωμές. Ε, δεν είναι δυνατόν παραδείγματος χάρη ε, όταν ε, κάποιες εταιρείες έχουν εταιρείε οι οποίες επεξεργάζονται τρόφιμα να δίνουν διάφορα μπόνους ανάλογα με τον χρόνο της ε, παράδοσης. Αλλά ε, βεβαίως ε, αν υπάρξει κάποια τέτοια ρύθμιση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι το οποίο να θέμει την εμπορική πρακτική σε μια χώρα να υπάρχουν και ανάλογες κυρώσεις. Δεν μπορεί, αν γίνει κάτι τέτοιο, να μείνει στο εθελοντικό επίπεδο. Βλέπουμε λοιπόν ότι στον ε, κλάδο των ε, τροφίμων δεν μπορούμε βεβαίως να καταργήσουμε την εθελοντική δέσμευση, αλλά όταν έχουμε κάποια κομμάτια τα οποία δεν συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία θα έπρεπε νομίζω να δούμε το θέμα. Το επόμενο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι ο διαχωρισμός μεταξύ δικαίου του ανταγωνισμού και της θέσης των παραγωγών. Προσπάθησα να δώσω κάποια παραδείγματα, να πω δηλαδή ότι θεωρούμε ότι όταν έχουμε οργανώσεις παραγωγών θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής νομική κατάσταση μεταξύ των δύο πλευρών. Παραδείγματος χάρη τώρα έχουμε τις πρώτες εξαιρέσεις στο πακέτο του γάλακτος και προσπαθούμε να επεκτείνουμε αυτές τις ρυθμίσεις και σε άλλους τομείς, στο κρέας, πάντα βασιζόμενοι σε ε, αναγνωρισμένες ενώσεις παραγωγών. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει σαφήνεια και διαφάνεια για το ποιοι ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές τις οποίες έχουμε. Με το θέμα λοιπόν της διαφάνειας της ε, αγοράς ε, έχουμε τους χάρη σας είπα ότι αναζητήσαμε παραδείγματα στις ίπα Θέλουμε λοιπόν να έχουμε περισσότερα και πιο γρήγορα από τα κατά την μέλη να λαμβάνουμε τα δεδομένα. Να αντιλαμβανόμαστε πού απαιτείται να αναλάβουμε δράση και βεβαίως να βοηθήσουμε την ε, αγορά και τους υπολογισμούς ε, του Food Euro, όπως λέγεται, και να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα στην ανάλυση κινδύνου. Και έρχομαι τώρα στην ανάλυση κινδύνου. Περνάμε λοιπόν, ναι, ε, χρειαζόμαστε ένα πακέτο εργαλείων διαχείρισης για το πώς θα μπορούν οι γεωργοί να διαχειριστούν ακριβώς αυτά, αυτούς τους ε, κινδύνους. Βεβαίω ε, είναι το ζήτημα του να αποφύγουν παραδείγματος χάρη την καταστροφή μιας σοδιάς, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και καλύτερη πληροφόρηση το που μπορεί να χρησιμοποιήσουν το χρηματοοικονομικό κλάδο για να προσφερθούν νέα εργαλεία στους γεωργούς για να αναλάβουν μεγαλύτερους ε, κινδύνους. Όλα αυτά βεβαίως ε, με τη βάση που προανέφερα. Και έρχομαι στην τελευταία εικόνα, τα συμβόλαια μελλοντική Εκπλήρωση. όπου έχουμε ακριβώς τους ε, νέους αυτούς κανόνες μετά την ε, δημοσιονομική κρίση όπου πρέπει να δούμε το τι θα γίνει με τα μέσα αυτά τα over the counter και το πιο ακριβώς είναι το όριο πρέπει να εξετάσουμε ακριβώς πού υπάρχει ακριβώς ε, ελλείψη ρευστότητας ε, και ισορροπίας ε, που υπάρχει ακριβώς ανάγκη για τέτοιες συμβάσεις. Παραδείγματος χάρη έχουμε την εικόνα στην αγορά των Δημητριακών που θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλους κλάδους και νομίζω μπορεί να αποτελέσει κάποια βάση για τέτοια προϊόντα over the counter και την επέκτασή τους. Νομίζω ο χρόνο δεν υπάρχει για τίποτα άλλο. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκίσεν. Όπως σας είπα, θα περάσουμε τώρα στα σχόλια της έκθεσης από τους καλεσμένους συμπειρογνώμονες. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάρτιν Μέριλτ από την ΚΟΠΑ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Επίτροπο και την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρωτοβουλία αυτή που ανέλαβαν προκειμένου να συσταθεί αυτή η δικαιωμάδα εργασία εργασίας για τις γεωργικές αγορές. Χαίρομαι ιδιαίτερος με αυτά που άκουσα και τα συμπεράσματα της Task Force αυτής, γιατί όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο την παραγωγή τροφίμων με δίκαιο τρόπο και την προστασία των γεωργών της Ευρώπης. Γιατί η γεωργία είναι σημαντικός κρίκος της τροφικής αλυσίδας. Χωρίς αυτούς δεν θα έχουμε τίποτα ε, για να παράγουμε, να μεταποιήσουμε, να εμπορευτούμε ή να καταναλώσουμε. Γι' αυτό η σημερινή συζήτηση στόχο έχει την προάσπιση της παραγωγής, της γεωργικής παραγωγής και της τροφικής αλυσίδας της Ευρώπης, ώστε να έχουμε ε, καλύτερα, πιο ποιοτικά και πιο φθηνά προϊόντα προς όφελος και των καταναλωτών αλλά και των παραγωγών. Επίσης, ε, τη στιγμή που πολλοί γεωργοί στην Ευρώπη έχουν υποστεί τεράστιες πιέσεις στην τροφική αλυσίδα και δεν αμείβονται δεόντως για την παραγωγή τους, γιατί αυτή είναι μια πραγματικότητα που την βλέπουμε καθημερινά σε πολλούς κλάδους παραγωγής. Θα πρέπει λοιπόν να δηλώσουμε πρώτα ξεκάθαρα ότι οι, Ευρω... Ευρωπαίοι Γεωργοί δεν λαμβάνουν με δίκαιο τρόπο το μερίδιό τους στην αλυσίδα αξιών της παραγωγής. Μάλιστα το ποσοστό έχει μειωθεί από 30% το 1995 στο 24% το 2005. Και αυτή η διαφορά ευνόησε περισσότερο άλλους κρίκους της τροφικής αλυσίδας και όχι τους γεωργούς. Δείχνουν οι στατιστικές ότι η προστιθέμενη αξία των γεωργών στην τροφική αλυσίδα ήταν μόνο 21% το 2011. Ενώ η προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας ήταν 28% και 51% ήταν για τους λιανέμπορους, για τις αλυσίδες διανομής και τις υπηρεσίες Οπότε από το ευρώ που ε, πληρώνει ο καταναλωτής, ένα πολύ μικρό μερίδιο παίρνει ο γεωργό και όλο και μικρότερο γίνεται αυτό το μερίδιο. Και μερικέ φορέ είναι μόνοι του οι γεωργοί στις διαπραγματεύσει απέναντι στις, ε, στους μεταποιητές και στις αλυσίδες διανομής που έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση. Ενώ οι γεωργοί είναι κατακαιρματισμένοι. Μάλιστα οι πέντε μεγαλύτεροι λιανέμποροι ε, είναι, έχουν ένα ποστό άνω το 60% φανταστείτε πόσο αδύναμη είναι η διαπραγματευτική θέση των γεωργών σε όλα αυτά. Του είναι το αποτέλεσμα για πολλούς γεωργούς είναι όλο, όσο και όλο και πιο παρατεταμένε ε, ε, περίοδοι αποπληρωμής. Έχουμε αναδρομικές αλλαγές σε συμβάσει, ε, αλλαγές τελευταία στιγμής, ακυρώσει τελευταία στιγμής. Και όλο και σημαντικότερη συμβολή τους στο κόστος. Όλα αυτά πλήττουν τους Γιώργους. Για παράδειγμα, ε, η μεγαλύτερη εταιρεία ελληνικού εμπορίου στην Ευρώπη είναι 7,5 φορές μεγαλύτερη από την μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής, την Friesland Campina. Βλέπετε ότι 7,5 φορές μεγαλύτερη είναι η ο έμπορος, ε, ε, ο λιανέμπορος γεωργικών προϊόντων από τον μεγαλύτερο παραγωγό γεωργικών προϊόντων. Και επίσης ε, ο κύκλος εργασιών του είναι πολύ μεγαλύτερος από τους 10 μεγαλύτερους γεωργικούς συνεταιρισμούς στην Ευρώπη. Βλέπετε τις τάξεις μεγέθους και πόσο εξασθενεί όλο και περισσότερο η διαπραγματευτική ισχύ των γεωργών εξαιτία αυτή τη συγκέντρωση των μεταποιητών και των αλυσίδων διανομή. Χαιρετίζουμε λοιπόν την έκθεση τη ειδική αυτή ομάδα εργασία για τι γεωργικέ αγορέ και περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε πώ θα εφαρμοστούν οι συστάσει του στην ευρωπαϊκή πολιτική στο μέλλον. Επίση, καλωσορίζουμε και την αναγνώριση ότι οι γεωργοί ε, έχουν περισσότερα κέρδη στις χώρες όπου είναι ενισχυμένη η συνεργασία τους και η οργάνωσή τους. Εδώ συμφωνούμε με την ε, ε, ομάδα εργασία θα πρέπει να προωθήσουμε τη, τους συνεταιρισμούς, τους γεωργικούς συνεταιρισμούς ε, και την οργάνωση των γεωργών σε οργανώσεις παραγωγών. Έτσι θα γίνουν πιο ανταγωνιστικοί οι γεωργοί, θα μειώσουν το κόστος τους και θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους ισχύ στην τροφική αλυσίδα υπάρχουν συνεταιρισμοί και οργανώσεις παραγωγών, αλλά θα πρέπει και ε, το δίκαιο ανταγωνισμού να εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου στους γεωργούς που οργανώνονται σε συνεταιρισμούς ή σε οργανώσεις παραγωγών. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις νομοθετικές διατάξεις ε, της ισχύουσας νομοθεσίας και να ενθαρρύνουμε τους ε, ε, γεωργούς να, να συσπηρωθούν και να συνενώσουν τις προσπάθειές τους ε, μέσω των συνεταιρισμών και των οργάνων, οργανώσεων παραγωγών. Μάλιστα, πολλά κρατημέλη ήδη έχουν υιοθετήσει εθνικές πρακτικές για να χαλιναγωγήσουν τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Γιατί κόπα κοζέκα είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν αυτές οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές μέσω όμως μιας ε, κοινοτικής πανευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα σέβεται και τις εθνικές ιδιαιτερότητες και τις ιδιαίτερες εθνικές δομές. Και γι' αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ισχυρό ρόλο των συνεταιρισμών και των ε, οργανώσεων παραγωγών και θα πρέπει να διαφυλαχθεί αυτό ο ισχυρό ρόλο στο μέλλον. Δεν θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου ο Γεωργό που ε, κατάφερε με επιτυχία να αυξήσει την διαπραγματευτική του ισχύ στην ε, τροφική αλυσίδα να αντιμετωπίζει περισσότερη γραφειοκρατία, περισσότερε νομοθετικέ διατάξει και αυξημένο κόστο. Επίση, η εύρυθμη λειτουργία τη εσωτερική αγορά έχει ζωτική σημασία και για να εξασφαλιστούν συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της τροφικής αλυσίδας και όλους τους κρίκους της αλυσίδας ε, εφοδιασμού, χρειαζόμαστε κοινοτική νομοθεσία για να χαλιναγωγήσουμε και να περιορίσουμε τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Και φυσικά θέλουμε και ανεξάρτητους φορείς ε, Εφαρμογή ε, των νομοθετικών διατάξεων για να αποκαταστήσουμε την ισορροπία στην τροφική αλυσίδα και να προστατεύσουμε καλύτερα του γεωργού. Έτσι, μια τέτοια εφαρμογή που θα εξασφαλίζεται από ανεξάρτητο τρίτο μέρο, ε, θα πρέπει να προβλέπει και δυνατότητα ανεξάρτητης διερεύνησης υποθέσεων και καταγγελιών για μη συμμόρφωση. Τα προβλήματά μας είναι ευρωπαϊκά, πανευρωπαϊκά και γι' αυτό και οι λύσεις θα πρέπει να είναι πανευρωπαϊκές. Και γι' αυτό οι σχετικές στάσεις της ομάδας εργασίας είναι πολύ σημαντικές. Στηρίζουμε αμέριστα ως Κοπακοζέκα τη χρήση των γραπτών συμβάσεων, γραπτών συμβολέων και αυτά θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά, τα γραπτά συμβόλαια. Επίσης ε, να γίνεται μια παρακολούθηση το επίπεδο των τιμών και να αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη. Έρχομαι στο διατάφτα. Είμαι βέβαιος ότι οι, Ευρωπαίοι καταναλωτές θέλουν τα προ... προϊόντα τους να τα παράγουν οι Ευρωπαίοι γεωργοί. Γι' αυτό και θα πρέπει να τους προστατεύσουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Είχαμε ακούσει πριν από λίγο τον πρόεδρο της ΚΟΠΑ Κοζέκα και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Γιώζεφ Πλάνκ, τον Γενικό Γραμματέα του Αυστριακού Γεωργικού Επιμελητηρίου. Παρακαλώ, πέντε λεπτά. Ε, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και εγώ την Κομισιόν για αυτή την έκθεση, την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναφερθεί σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα για την γεωργία, γιατί ο ρόλος της συμμετοχής των αγροτών στην αλυσίδα της δημιουργίας αξίας είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να φέρω κάποιες πτυχές από τη δική μου τη χώρα. Αφενός έχουμε μια πάρα πολύ έντονη συγκέντρωση του τομέα όσον αφορά τις ε, επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν ε, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα κτλ. Και στην Αυστρία παρατηρούμε ότι επίσης τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα καλύπτουν και το 86% ε, της αγοράς των τροφίμων. Οπότε βλέπετε ότι παίζουν και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και οι αγοραστές των γεωργικών προϊόντων. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμοστούν κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα ο ρόλος ε, του να μπορούν οι αγρότες ε, να κοιτάνε ως ε, ίση τις επιχειρήσεις εμπορίας τροφίμων και εδώ πέρα θα έπρεπε ακριβώς να δούμε το θέμα της αγοράς, ε, της εμπορίας ε, τροφίμων. Το συζητάμε συχνά. Ποια είναι, παραδείγματο χάρη, η δεσπόζουσα θέση σε μια τέτοια αγορά, ποια είναι η θέση των αγροτών. Και αυτό οπωσδήποτε δεν μπορεί να συνεχιστεί ως κατάσταση και στο μέλλον και όπως είπαμε χρειάζονται ξεκάθαρες ε, προοπτικές και θα πρέπει ξεκάθαρα να υπάρξει μια κατάσταση η οποία δεν θα έρχεται σε σύγκρουση με το δίκαιο του ανταγωνισμού για να μπορούμε έτσι να συνομιλούμε ως ίση και για τιμές, προθεσμίες, προϊόντα και στο επίπεδο των συμβάσεων όπως αναφέρατε με τους ανθρώπους οι οποίοι αγοράζουν τα προϊόντα μας γιατί αυτή τη στιγμή μας ρίχνουν ένα συμβόλαιο στο τραπέζι και αυτό είναι και άμα θέλουμε. Ε, δεν υπάρχει λοιπόν και η ανάλογη δύναμη διαπραγματευτική από πλευράς ε, των ε, ενώσεων αγροτών οι οποίοι βρίσκονται σε μια θέση όπου είναι στο κέντρο ενός και συμπιέζονται και από τις δύο πλευρές. Μετά περνάμε και με αυτό το θέμα στις αθέμητες εμπορικές πρακτικές που προκύπτουν συχνά και βεβαίως ε, είναι προφανές ότι ε, γίνονται κάτω από το τραπέζι και πρέπει να γνωστοποιηθούν ε, πολύ περισσότερο. Κοιτάμε, παραδείγματος και άλλα ζητήματα. Αναφέρθηκε και το ζήτημα της βιωσιμότητας της παραγωγής, όπου απαιτούνται πάρα πολλά μέτρα. Βλέπουμε εδώ πέρα πως τα παραδοσιακά μέσα ε, είναι πάρα πολύ στοχευμένα και δεν είναι πάρα πολύ απλό να ενσωματώσουμε εδώ πέρα νέα μέσα για την διασφάλιση απέναντι στους κινδύνους. Εσείς μιλήστε παραδείγματο χάρη για την αντασφάλιση. Και βεβαίω υπάρχουν ε, ζητήματα τα οποία μας προβληματίζουν και θα πρέπει να δούμε και τα παραδοσιακά μέσα για την διασφάλιση κινδύνου για την ασφάλιση της σοδιάς, δηλαδή αυτά τα οποία είχαμε παραδοσιακά τόσα χρόνια. Επιπλέον, έχουμε τις σκέψεις που έρχονται από την Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, παραδείγματος χάρη, όταν μιλάμε για τις αγορές της βιοενέργειας, των βιοκαυσίμων. Εκεί πέρα βλέπουμε ότι έχουμε τις εξελίξεις αυτών των ε, τομέα, κάτι το οποίο επίσης θα αποτελέσει ένα σημαντικό κριτήριο και μια μεγάλη πρόκληση για το μέλλον, για την αηφορία, για την κλιματική πολιτική, για το περιβάλλον, κάτι το οποίο βέβαια μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την συνεργασία της ε, Γεωργίας. Και ένα άλλο σημείο στο οποίο θα θέλαμε να εστιάσουμε, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, πάρα πολλούς ε, κανόνες, ε, τους οποίους σκεφτόμαστε. Συχνά είναι κανόνες οι οποίοι βεβαίως μπορούν να εφαρμοστούν από μεγάλες εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις, αλλά είναι κάτι το οποίο πραγματικά πνίγει τους μικρούς αγρότες οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν και έχουν φτάσει στα όρια τους, οικογενειακές επιχειρήσεις ε, και στην γεωργία πραγματικά έχουν φτάσει στο όριο τους. Είτε μιλάμε για διατάξεις ποιότητας, ε, πιστοποίησης, όλα αυτά μπαίνουν εκεί πέρα. Όταν τα πράγματα γίνονται υπερβολικά, αυτοί οι οποίοι πλήττονται είναι οι πιο μικροί και οι πιο αδύναμοι. Έχουμε λοιπόν παγκόσμιες αγορές, οπότε θα έπρεπε και οι κανόνες μας να ισχύουν τουλάχιστον για όλους όσους είναι στην ε, αγορά μας. Έτσι, αυτό νομίζω είναι το ελάχιστο. Σας ευχαριστώ και τώρα λόγω στον κύριο Μπέρι Χρέιμοντ, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Γεωργών του Ηνωμένου Βασίλειου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Πίτροφε Χόγκαν, Δόκτωρ Κίσεν, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για αυτή την ευκαιρία να πω μερικά λόγια σήμερα. Ευχαριστώ και σας Επίτροπε Χόγκαν που προωθήσατε αυτή την έκθεση και ευχαριστώ και την ομάδα Κρούσης για την εκπόνηση αυτή της πολύ καλής εκθέσεως. Σαν εκπρόσωπος της ΚΟΠΑ στο Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την Εύρεθμη Λειτουργία της Αρισίδας αποδεισμού τροφίμου και πρόεδρος της Εθνικής Ενώσεως ε, Γεωργών Αγγλίας και Ουαλίας. Εκπροσωπούμε πολλά μέλη και καλωσορίζω την έκθεση της ε, ομάδας κρούσης και τις συστάσεις που περιέχει. Και υποστηρίζω τις απόψεις του κ. Μάρτιν και του κ. Πλάνκ στα δεξιά μου. Η ομάδα κρούσης εξαπώνησε ένα έγγραφο. Πρέπει αυτό να απαιτήσει από τους διαμορφώντες την πολιτική να λάβουν πρωτοβουλίε για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, τα αφισβήτητα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί στην τροφιμική αλυσίδα. Σήμερα θα ήθελα να τονίσω έναν συγκεκριμένο τομέα. Πιστεύω ότι εκεί αμέσως μπορούμε να κάνουμε βήματα σε αυτόν τον τομέα για να κάνουμε τη διαφορά. Θα επικεντρωθώ επί του σημαντικού ζητήματος της διαφάνειας της αγοράς. Είναι θετικότατο ότι η ομάδα κρούσης αναγνώρισε την ανάγκη να υπάρχει σωστή ενημέρωση της τιμές για να βελτιωθεί η διαφάνεια ε, της αγοράς. Κόπερ και NFU ζητήσαμε συχνά να καλυφθούν οι μαύρες τρύπες που υπάρχουν όσον αυτά τα στοιχεία για την αγορά και για τους φορείς μεταποίησης. Διότι έτσι δεν δημιουργείται εμπιστοσύνη, μειώνεται συνεργασία και δεν αναπτύσσονται τα σωστά εργαλεία διαχείριση των κινδύνων της αγοράς. Πολλοί αναφέρθηκαν ότι χρειάζεται προσέγγιση με στόχο την αγορά όσον αφορά τη διαχείριση του κινδύνου. Για να αλλάξει η προσέγγιση πρέπει να έχουμε τα σωστά θεμέλια. Χρειάζονται σωστές συνθήκες λειτουργίας για τον τομέα της γεωργίας. Ακριβώς, για αυτό το λόγο, η υποχρεωτική υποβολή αναφορών στις τιμές πρέπει να εφαρμοστεί. Πρέπει να είναι υποχρεωτική αυτή διότι δεν υπάρχουν εθελοντικά μέσα που θα εξασφαλίζουν αξιοπιστία, ακρίβεια και έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων πληροφοριών για την υποστήριξη λύσεων που βασίζονται στην αγορά όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων. Σωστά, η Task Force αναφέρεται στην ανισορροπία μεταξύ ε, των διαφόρων τομέων της τροφιμικής αλυσίδας. Τον έφερε ο κ. Μάρτιν Μέριλ. Αυτό μαζί με τις διαφορές που υπάρχουν αφορά το σχετισμό δυνάμων μεταξύ μεταποιητών και γεωργών και ελιανοπολιτών, αυτό δείχνει ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού σε τρόφιμα. Η υποχρεωτική υποβολή των τιμών θα βοηθήσει να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη και να βελτιώσουμε τις σχέσεις μεταξύ γεωργών και όλων των φορέων της τροφιμικής αλυσίδας. Σχετικά με αυτό, η θέσπιση συστήματος υποβολής των τιμών είναι βασική συνιστόσα για να πετύχουμε και αυτά που ζητούν οι άλλες συστάσεις της ομάδας κρούσης. Είτε εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου ή για τις ε, διάφορες συμβάσεις μελλοντικής απόδοσης, ε, καλύτερη συνεργασία μεταξύ παραγωγών, καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση κλπ. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που παρατίθενται από την ομάδα κρούσης. Τον είπα όσον αφορά τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Ισπανία, όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις τιμές. Και αυτή η διαφάνεια βελτίωσε την εμπιστοσύνη στον τομέα. Και χαίρομαι που το τονίσατε, κύριε Γκίσεντ. Καλωσορίζω τη δημιουργία του παρατηρητηρίου για την αγορά, παρατηρητήριου για την αγορά, για να συλλέγονται χρήσιμα στοιχεία. Όμως, κατεπηγόντως, θα πρέπει να ελέγχονται οι πληροφορίες που παρέχονται όσον αφορά τα παρατηρητήρια του τομέα του γάλακτος. Αυτό είναι χρήσιμο για την έρευνα και τη διαμόρφωση πολιτικής. Δεν βοηθά όμως πολύ τις επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους τους άμεσους. Υπάρχει χρονική στέρηση στην υποβολή των τιμών. Και η ομαδοποίηση των στοιχείων χρειάζεται χρόνο. Δεν είναι τυποποιημένα τα στοιχεία. Άρα οι αναφερόμενες τιμές πολύ συχνά είναι απειρχιωμένες. Δεν αντικατοπτρίζουν την τοπική δυναμική, της ανάγκης των επιχειρήσεων. Σωστά είπε όμως η Task Force ότι υπάρχουν τεχνικές λύσεις. Αυτές μπορούν να δώσουν κατάλληλες πληροφορίες που απαιτούνται έγκαιρα και με ευθυνό τρόπο. Κλείνοντας, θέλουμε να είναι δυναμικό ο τομέα. Να υπάρχει σωστή συνεργασία των πτυχών για την μετώπιση των κινδύνων. Να υπάρχει ανταπόκριση στις τάσεις των καταναλωτών. Όμως, η συνεργασία προέρχεται από εμπιστοσύνη και εμπιστοσύνη από ανοιχτή προσέγγιση. Η υποχρεωτική υποβολή αναφορών όσον αφορά τι τιμέ είναι κρίσιμο άμεσο βήμα πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε το άνοιγμα. Για να προωθήσουμε καλύτερη πρόβλεψη τη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά και να αποκατασταθεί, να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνη στην αγορά. Σα ευχαριστούμε θερμά. Και περνάμε στον τελευταίο μα καλεσμένο, τον καθηγητή Πένιγκ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαίρω την Task Force για την έκθεση. Θα εστιαστώ σήμερα επί δύο κεφαλαίων. Για τη διαχείριση του κινδύνου και για τα συμβα... συμβάσεις μελλοντικών αποδόσεων. Θα χρησιμοποιήσω διάφορα στοιχεία από την έκθεση, παραθέσεις από το κείμενο, με και κλειμένους χαρακτήρες και εντό εισαγωγικών. Η διαχείριση του κινδύνου αντιμετωπίζει το κόστος του κεφαλαίου. Η πρόκληση για τους γεωργούς είναι το κόστος του κεφαλαίου. Είναι πάρα πολύ υψηλό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μόνος τρόπος να χρησιμοποιήσουμε το κόστος κεφαλαίου για τη διαχείριση του κινδύνου αν έχουν πολύ ψηλό κόστος κεφαλαίου δεν θα μπορούμε να καινοτομήσουμε. Γι' αυτό τονίζω το κόστος κεφαλαίου σημαντικό παράγοντα. Η διαχείριση του κινδύνου μέσω μειώσεως της μεταβολής του κόστους αυτού είναι η δύναμη για να μειώσουμε την, το κόστος κεφαλαίου. Η έκθεση εντοπίζει ότι υπάρχει μεγάλη τερογένεια στον αφορά τους κινδύνους. Και θα ήθελα να τονίσω ότι η ετερογένεια υπάρχει όσον αφορά και τις τάσεις εναντί του κινδύνου και την αντίληψη του κινδύνου πλευράς γεωργών. Αυτό συνεπάγεται ότι η διαχείριση του κινδύνου, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε επίπεδο εκμετάλλευσης. Ο γεωργός πρέπει να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο σε συνάρτηση ε, με την έκθεσή του στον κίνδυνο. Τώρα, Ποιο είναι ο ρόλο αγορά μελλοντικών αποδόσεων, συμβάσεων μελλοντικών αποδόσεων. Δεν θα μιλήσω για το θέμα τη προστασία αυτών, αλλά την κάλυψη των τιμών. Και άλλα μέλη είπαν ότι η ποιότητα των στοιχείων είναι σημαντικότατη. Τι εννοώ. Αν οι τιμέ βασίζονται αποκλειστικά στι συναλλαγέ. Πολλέ τιμέ που χρησιμοποιούμε στι Βρυξέλλε δεν βασίζονται επί πραγματικών συναλλαγών. Κάτι άλλο που ανέφερε ο κ. Ρέιμοντ ε, είναι η χρονική στέρηση. Οι τιμές βασίζονται σε πραγματικές συναλλαγές. Χρειάζεται σωστός χρονικός συντονισμός. Ε, έγκαιρη μεταβίβαση των τιμών. Αυτό χρειάζεται ο Γιώργος και χρειάζονται και ισότιμες συνθήκες. Ε, να μπορούν όλοι να γνωρίζουν τις τιμές. Αυτό βοηθάει και τους Γιωργούς. Θα μπορούν να αξιολογήσουν τις συμβασιακές σχέσεις που υπάρχουν. Στην έκθεση αναφέρεται το θέμα των συμβάσεων. Σαν γεωργό θα πρέπει να αξιολογήσω κατά πόσο η σύμβαση που μου προσφέρεται είναι λογική ή όχι. Και σαν γεωργό πρέπει να δω και ποια θα είναι η μελλοντική τιμή. Οπότε το θέμα των μελλοντικών αποδόσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ για να λάβω μια θέση στην αγορά. Βοηθάω όμως για να καταλάβω πώς μπορώ να ερμηνεύσω τη διαμόρφωση των τιμών. Δύο συνιστώσεις έχουμε εδώ. Που είναι κρισίμου σημασία όταν μιλάμε για το hedging. Συνιστώσεις που διαμορφώνται στην πολιτική και οι γεωργοί θα πρέπει να αντιληφθούν. Η αποτελεσματικότητα της προστασίας του hedging και η βελτιοποίηση των ποσοστών. Θα πρέπει να μειώνεται ο κίνδυνος όσον αφορά των συμβάσεων μελλοντικής απόδοσης, διότι οι συμβάσεις μελλοντικών αποδόσεων ε, εισάγουν κινδύνους. Πρέπει να προσμετρήσουμε αυτούς και να αξιολογήσουμε πώς μπορούν αυτές οι συμβάσεις να βοηθήσουν την αντιμετώπιση των κινδύνων. Άρα θα πρέπει να εντοπίσουμε τα βέλτιστα ποσοστά προστασίας. Είναι του hedging. Είναι βασικές παράμετροι που πρέπει να γνωρίζουν οι γεωργοί και οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι, να κατανοούν. Αν μπορέσουν να το κάνουν αυτό και αυτοί που διαμορφώνουν την πολιτική και οι γεωργοί, τότε είμαι πεπισμένος ότι οι γεωργοί μπορούν να αυξήσουν την αντοχή τους στην οικονομική εστιαζόμαστε συχνά επί των επιπέδων των τιμών, το κατανοώ. Πιο σημαντικό είναι να βλέπουμε και πώς μεταβάλλονται οι τιμές, αν είναι ευμετάβλητες. Όπως έδειξα και στην πρώτη μου διαφάνεια, η μεταβολή των τιμών και η διαχείριση της μεταβολής των τιμών μειώνει το κόστος του κεφαλαίου και αυξάνει την αξία της εκμετάλλευσης. Άρα εξασφαλίζεται ότι μπορεί να καινοτομεί ο Γιώργος αδιαμφισβήτητα αποφασιστικός παράγων για επιτυχή γεωργία είναι η δυνατότητα του γεωργού να χειρίζεται το κίνδυνο. Να το συσχετίσουμε με μια έρευνα που πραγματοποίησαμε. Παρακολουθήσαμε επί 10 χρόνια εκμεταλλεύσεις. Και τι κάναμε. Τις ταξινομήσαμε ανάλογα με την επίδοσή τους. Ποιο ήταν το ενδιαφέρον. Ότι βλέπουμε κάποιους γεωργούς που πάντα τα πηγαίνουν καλύτερα. Αποδίδουν καλύτερα και δεν σχετίζεται με το μέγεθος εκμετάλλευσης αυτό, σχετίζεται με τη διαχείριση του κινδύνου. Τι δυνατότητα έχουν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Η δυνατότητα εκτέλεσης ενός σχεδίου διαχείρισης του κινδύνου της αγοράς είναι αποφασιστική σημασία για την επιτυχία του γεωργού, αν αποδίδει καλά η επιχείρησή του. Τι πρέπει να κάνουμε. Χρειαζόμαστε ένα δικό χάρτη. Νομίζω ότι η ομάδα Κρούσης έκανε υπέροχη δουλειά ενετόπισε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Τώρα θα πρέπει να τα λύσουμε. Ποιο είναι το ενδιαφέρον. Η Task Force αναφέρεται συχνά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά η γνώση για διαχείριση κινδύνου και τις συμβάσεις μελλοντικής απόδοσης είναι εδώ. Οι Αμερικανοί έρχονται στην Ευρώπη για να αποκτήσουν τεχνογνωσία για αυτά. Εκεί που είπα μας ξεπερνούν είναι στη χρήση της γνώσεως και της άμεσης εφαρμογής αυτής σε επίπεδο εκμετάλλευσης. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι χρειαζόμαστε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές. Το προηγούμενο μέλος του πάνελ το εντόπισε αυτό. Ότι χρειάζεται αναφορά των τιμών και να αυξηθεί διαφάνεια στην αγορά. Αν τα εφαρμόσουμε όλα αυτά, θα είμαστε σε καλή φόρμα και θα καταφέρουμε να έχουμε ανθεκτικές, πραγματικά ανθεκτικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα στους συντονιστέ. Δύο λεπτό ο καθένας. Ο κύριος Αλμπερτές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους με υγεία και επαγγελματική επιτυχία. Λοιπόν, θα δώσω όμως αμέσως τον ε, λόγο στον ε, συνάδελφο γιατί θα πρέπει να φύγει από την αίθουσα. Κύριος Νταντά, ευχαριστώ Άλμπερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, μέλη της ε, ειδική Ομάδας Εργασίας, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Άλμπερ Ντες που μου παραχώρησε τη θέση του γιατί πρέπει να σπεύσω σε άλλη συνεδρίαση. Ε, έχουμε μια σοβούσα γεωρική κρίση και η Επιτροπή για τις Γεωργικές Αγορές και η Ειδική Ομάδα Εργασίας ε, συστήθηκε ακριβώς για αυτό το λόγο και είναι αξιοσημείωτο το έργο και πολύ αξιόλογό της. Γιατί ε, ενισχύει και θα τη συζήτηση μεταξύ των διαφόρων φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού υποβάλλεται στάσεις για τη σχέση μεταξύ των διαφόρων παραγόντων τη αλυσίδα αναφοδιασμού και οι προτάσεις σα επίσης, οι ε, νομοθετικέ, ε, είναι πολύ σημαντικέ. Έχουμε και τη συνάδουμε τη, τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα πρόσφατα συμπεράσματα του Γεωργικού Συμβουλίου. Και μάλιστα ένας υπάλληλο Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ασχολείται ιδιαίτερα με τα θέματα αυτά και θα καταλάβει ποιον εννοώ, είπε ότι ο πλανήτης ε, ευθυγραμμίζεται, γι' αυτό και η ευθύνη μας ε, για ανάληψη δράσης γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Ο γεωρικός ε, πληθυσμός περιμένει άμεσες απαντήσεις για να, για να αποκατασταθεί η ισορροπία στην ταφική αλυσίδα, να, ξανα... να αναθεωρήσουμε τις οικονομικές σχέσεις και να θαρρύνουμε τη δραστηριότητά της. Και χαίρομαι για το θάρρος που έδειξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πρωτοστατήσει αυτή τη συζήτηση και για το δίκαιο ανταγωνισμό, με κοινή πρωτοβουλία του Συμβουλίου και της Επιτροπής προκειμένου να υποβληθούν φιλόδοξες προτάσεις και θα πρέπει να είναι γίνουν αντιληπτέ από όλου του παράγοντε. Και μάλιστα το δίκαιο ανταγωνισμού για τα γεωργικά θέματα θα πρέπει να απλουστευτεί και να διευκρινιστεί. Και ελπίζω να συνεργαστούμε στενά στο εγγύ μέλλον για το θέμα αυτό, να απλουστεύσουμε το δίκαιο ανταγωνισμού. Και μάλιστα ε, η παρουσία τη Επιτρόπου Φαριστάκη 28 Φεβρουαρίου στην ακρόαση που θα έχουμε θα είναι σημαντικό βήμα πρόοδου. Χαίρομαι για το κουράγιο που δείχνουμε και την πρόθεση τη συζήτηση για την διαφάνεια τη αλυσίδα και την καταπολέμηση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Η προστιθέμενη αξία θα πρέπει να κατανέμεται ισορροπημένα μεταξύ των διαφορών κρίκων τη τροφική αλυσίδα και όχι να αποβαίνει βάρο των γεωργών. Όλα αυτά θα πρέπει να καθοδηγήσουν το έργο μα και για, την, για τον, το πακέτο νομοθετικό και για τη μεταρρύθμιση της κοινή ζωρική πολιτικής. Θέλουμε πιο διαφανείς λύσεις για μια πιο ισορροπημένη και διαφανή τροφική αλυσίδα, έστω και αν αυτό αυξήσει κάπως την τιμή καταναλωτή. Γιατί έχουμε και άμεσε ενισχύσει που κάθε 5-6 χρόνια τι αναδιαπραγματευόμαστε, θα μπορούσαμε μέχρι το δεύτερο, από το δεύτερο πυλώνα να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα θέματα, γιατί έχουμε τακτικέ διαπραγματεύσει γι' αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θα επιβαρύνει τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Κάτι που είναι πολύ θετικό. Ενώ ο αντίκτυπο θα είναι πολύ καλύτερο και σημαντικότερο για την αύξηση τη ανθεκτικότητα του γεωργικού κλάδου. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γιλέρα. Ε, μια και απουσιάζει ο κύριος Δεκάστρο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Καλή χρονιά σε όλους εύχομαι και ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του συντονιστή μας, του Παύλου Τεκάστρο, που δυστυχώς ε, δεν μπόρεσε να έρθει εγκαίρος. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την ομάδα εργασίας για την πολύ αξιόλογη και ενδιαφέρουσα έκθεση και συμπεράσματα που υπέβαλε. Όπως είπε και ο κύριος Νταντάν, ε, έχουμε αναφυσβήτα πολλά κοινά σημεία μεταξύ της έκθεσης ομάδας εργασίας και της ε, έκθεσης της Επιτροπής Γεωργίας και το είπε και ο κύριος Γκίζεν ότι τα εθελοντικά μέτρα είναι θετικά μένα αλλά δεν αρκούν. Θα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις για να παταχθούν οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές και να είναι δεσμευτικές αυτές οι προτάσεις, να μην περιορίζονται μόνο σε εθελοντικά μέτρα. Επίσης, να ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική ισχύ των γεωργών. Ε, και στη Σοσιαλιστική Ομάδα θα έρθει ο κ. Επίτροπο του Ιανουάριο, για να συζητήσουμε ακριβώ πώ θα αποκαταστήσουμε την ισορροπία τη τροφική αλυσίδα και θα ενισχύσουμε την διαπραγματευτική ισχύ των γεωργών. Είχαμε ενδιαφέρουσε εθνικέ πρωτοβουλίε στην Ισπανία, για παράδειγμα, με το σχετικό νόμο για την τροφική αλυσίδα. Αλλά έχουμε ενιαία αγορά και μπορεί μεν κάποιε κυβερνήσει να έχουν ε, αγαθέ προθέσει και να υποβάλουν κάποια μέτρα, αλλά δεν θα έχουμε θετικό αντίκτυπο σε όλε τι τιμές. Γιατί είχαμε κρίσεις όχι μόνο στο γαλακτοκομικό τομέα και σε άλλους, παρά τις θετικές ενέργειες μεμονωμένων κυβερνήσεων. Γι' αυτό και τα συμπεράσματα τη ομάδα εργασία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Θέλουμε και ασφάλεια δικαίου στο δίκαιο ανταγωνισμού, γιατί υπάρχουν πολλέ αμφιβολίε και θα πρέπει να τι διευκρινίσουμε και να διασκεδάσουμε τι αμφιβολίε. Να διαφυλάξουμε το σημαντικό ρόλο των συντενετερισμών και των, ε, ε, των οργανώσεων παραγωγών. Και η έννοια του συνεταιρισμού νομική ε, προσωπικότητα και οντότητα είναι πολύ σημαντική, και θα πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Έχουμε μια συγκεκριμένη ερώτηση, κυρία Γκίζεν. Ποιο θεωρείτε ότι είναι ο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι διακλαδικέ ε, διαπαγγελματικέ οργανώσει ε, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί δεν το αναφέρατε. Έχουμε κάποιε περιφερειακέ εθνικέ διατάξει, αλλά ίσω ήταν σκόπιμο να έχουμε και ευρωπαϊκέ διατάξει για τι διαπαγγελματικέ οργανώσει. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά κύριε Γκίζεν. Αυτά ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ ο κύριος Χαϊτεμά από τους Φιλελεύθερους. Eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και για τις ε, παρουσιάσεις. Συγχαρητήρια για την έκθεση. Είναι πολύ συγκεκριμένη, σαφής, ξεκάθαρη και μας δείχνει το τι πρέπει ακριβώς να γίνει δύο πράγματα από μένα που είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτα απ' όλα η νομοθεσία η οποία έχει περισσότερες προβλέψεις για την ε, συνεργασία και τις ομάδες των παραγωγών και για τις αγορές γιατί βεβαίως η αγορά δεν ε, συνεργάζεται ε, με, δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο παντού. Παραδείγματο χάρη, οι αγοραστέ των προϊόντων συνεργάζονται, αλλά δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο παραγωγή για τον απλούστο λόγο ότι δεν έχουν ε, τα μέσα να πληρώσουν νομικού ή την απαραίτητη εμπειρία. Θα πρέπει εδώ πέρα λοιπόν να δούμε αυτό το θέμα. Το ζήτημα και το ερώτημά μου είναι το εξή. Όταν μιλάμε για το δίκαιο του ανταγωνισμού. Πού θα θέλατε να ρίξει το βάρος του και να δώσει σημασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μιλήσατε για μια ένταση μεταξύ Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Ανταγωνισμού. Πώς θα πρέπει να συνεργαστούν για να έχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Δεύτερον, διαχείριση κινδύνου και μέσα διαχείριση του κινδύνου θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε στο περιβάλλον της ε, παγκοσμιοποίησης το πώς θα μπορέσουν να διασφαλιστούν ε, περισσότερο οι αγρότες και είναι σημαντικό να έχουμε κάποια συγκεκριμένα εργαλεία, κάποια μέσα για να μπορούμε να καλυφθούμε από, συνθήκου, από κινδύνους ε, καιρού, παραδείγματος χάρη, η διακύμανσης τιμών. Υπάρχουν κάποια μέσα στην Ολλανδία. Δυστυχώς η συμμετοχή των αγροτών είναι πάρα πολύ χαμηλή, αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη υπάρχουν... Δέκα κράτη-μέλη που εκμεταλλεύονται τα κονδύλια του δεύτερου πυλώνα για τις ε, γεωργικές ε, ασφαλίσεις και για την σταθερότητα του εισοδήματος. Πώς μπορούμε λοιπόν να φροντίσουμε να υπάρξει ακριβώς μεγαλύτερη υιοθέτηση αυτών των ε, μέσων του δεύτερου πυλώνα. Θα πρέπει να έχουμε έναν οδικό χάρτη όπως μας πρότεινε ο συνάδελφός σας. Θα πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τέλος, πριν χτυπήσει το σφυράκι ο πρόεδρος, τι μπορούμε να μάθουμε από τις ΗΠΑ Ακούσαμε τον κύριο Πένινγκ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ περισσότερη γνώση αλλά δεν την χρησιμοποιεί. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο κατά την άποψή μου που να δείχνει ότι πρέπει να φρονούμε ότι το 2017 θα οδηγήσει μεγαλύτερη σταθερότητα των τιμών για τους γεωργούς από τα τελευταία χρόνια. Όλα τα σημάδια δείχνουν ότι οι γεωργοί θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις των τιμών και μεγαλύτερους κλειδονισμούς στις τιμές, βλέποντας τον αντίκτυπο του Brexit και των άλλων διεθνών γεγονότων και πολιτικών γεγονότων που θα λάβουν χώρα πιθανότατα κατά τη διάρκεια του 12 μήνου. Θα υπάρξουν αλλαγές. Θα υπάρχουν κλειδονισμοί όσον αφορά τις τιμές. όσον αφορά τα γεωργικά τρόφιμα. Το θέμα είναι ποιος θα απορροφήσει αυτά τα πλήγματα. Κάθε κρίση τιμών που συνέβη τα τελευταία χρόνια μας έδειχνε ότι οι γεωργοί τελικά δέχονται το πλήγμα των κλειδονισμών. Εκτός αν εμείς, όταν λέω εμείς, ενώ συλλογικά εμείς κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμείς το Κοινοβούλιο, αν όλοι πούμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δημιουργούν την αλυσίδα για τα τρόφιμά μας από την εκμετάλλευση μέχρι τα στο πιάτο μας. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ε, δίκαιη διανομή όσον αφορά τα κέρδη και όχι μόνο αυτό, αλλά και οι απώλειες πρέπει να μοιράζονται δίκαια. Ανεξάρτητα από αυτά που ακούω από τις οργανώσεις των γεωργών είτε εκπροσωπούν τη γαλακτοδομία, το χείριο κρέας, το βόλιο κρέας, όταν μου λένε ότι οι τιμές τους μειώθηκαν μέχρι και 50% σε κάποιες περιπτώσεις και πάω στην υπεραγορά μου, στην τοπική, δεν βλέπω μείωση 50% των τιμών. Αν δεν αντιμετωπίσουμε τους μεταποιητές και τους λιανοπολιτές που κρατούν ομήρους τους ε, γεωργούς μας όσον αφορά τις τιμές, εάν δεν το κάνουμε αυτό δεν θα λύσουμε τα προβλήματα. Πρέπει να ξεχάσουμε εθελοντικούς κώδικες για μεταποιητές και λιανοπολιτές. Πρέπει να του αντιμετωπίσουμε στεναρά, να μην τους επιτρέπουμε να πολλούν τα γεωργικά προϊόντα σε τιμή κάτω του κόστους και να πιέζουν τους παραγωγούς μας. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά και από μένα συνεχίζουμε την ίδια συζήτηση που έχουμε εδώ και χρόνια και την ίδια λύση. Αυτό το οποίο δεν βλέπουμε είναι πολιτική δράση, συγκεκριμένες προτάσεις. Πού είναι εδώ πέρα ε, ο κλάδος του ανταγωνισμού να μας πει τι επιτρέπεται και τι όχι. Κάνουμε τη δικιά μας την εσωτερική συζήτηση όπου συμφωνούμε αλλά δεν προχωράμε καθόλου και αφήσατε κάποια ε, εργαλεία εκτός. Μιλήσατε για τιμές, δεν μιλήσατε για ποσότητες. Ε, το είδαμε αυτό στον τομέα του γάλακτος. Όταν υπάρχει υπερβολική παραγωγή, μπορείτε να παρατηρείτε τις τιμές όσο θέλετε, αλλά πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία στην αγορά. Ε, μπορούμε να μειώσουμε λοιπόν την προσφορά και αυτομάτως ανεβαίνουν οι τιμές. Μπορούμε να το επαναλάβουμε αυτό το φαινόμενο, το, το γιογιό, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να προσαρμοστούν οι ποσότητες στη ζήτηση. Έτσι θα αποκτήσουν τη δύναμη οι γεωργοί. Για την πρόταση για όμπουτσμαν. καλή, αλλά τελικά θα καταλήξει να είναι ένα σε κάθε χώρα. Η λύση σας που προτάθηκε είναι να πάνε στα χρηματιστήρια και στις προθεσμιακές αγορές οι οι αγρότες. Ναι, ναι, αυτό μπορεί να χρειάζονταν ε, λίγη ακόμα κερδοσκόπη. Δεν ξέρω τώρα ειλικρινά με τόσο ευπαθή και ευαίσθητα προϊόντα εάν μπορούν να πάνε σε τέτοιες αγορές. Γιατί είναι άλλα τα ζημητριακά και άλλα τα, τα ευπαθή. Δηλαδή πάντα παρουσιάζεται αυτή η πρόταση αλλά δεν στέκει για πολλούς κλάδους γεωργίας. Ενίσχυση των παραγών, ναι ωραία, και συνεταιρισμοί. Να σας πενθυμίσω εδώ πέρα πως ε, ε, τελικά και οι συνεταιρισμοί δεν χρησιμεύουν σε τίποτα αν δεν έχουν δύναμη. Αυτό αποδείχθηκε στη μεγάλη κρίση του γάλακτος στη Γερμανία. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουν όντως δύναμη οι συνεταιρισμοί και βλέπουμε ακριβώς ε, το πρόβλημα και με την αγορά και το πόσο αυτό περιορίστηκε η νομοθεσία στον τομέα του γάλακτος. Επίσης, όταν μιλάμε και για τα ποιοτικά προϊόντα και στο γάλα και εκεί πέρα νομίζω μπορούμε να επηρεάσουμε έτσι την αγορά. Νομίζω προς τα εκεί θα πρέπει να πάει η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συζητούμε τις, την Task Force και την έκθεσή της για τις αγροτικές ε, αγορές αλλά ίσως μπαίνει σε κάποιους τομείς όπου δεν θα έπρεπε να μπαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα για το εμπορικό δίκαιο, Φερρυπίν, και κάποιες συστάσεις της εκθέσεως θα πρέπει να ενεργοποιηθούν τι ούτω τρόπος. Δεν έχει τη δικαιοδοσία όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά το θέμα των εξαιρέσεων από το φόρο εισοδήματο κλπ. Φορολόγηση αυτά είναι αρμοδιότητα κρατών μελών και δεν μπορεί να επηρεάζεται από εμά. Κάτι για την υποβολή αναφορών για τις τιμές, για την ενημέρωση για τις τιμές. Ε, για το ζαχαρότευτο γνωρίζουν τι παίρνουν οι γεωργοί, για το σίτο, για τα αυγά κλπ. Αφού το σκάλισαν οι δημοσιογράφοι, ξέρει ο κόσμος τις τιμές. Στην άλλη άκρη του κλίμα, του, της κλίμακας όλοι γνωρίζουν ποια είναι η τιμή στις υπεραγορές των τροφίμων. Θέλω κανένα δύο κάποια παραδείγματα τον κύριο Ρήμοντ. θέλει πόσο παίρνει ο μεταποιητής από την υπεραγορά. Αρκετή ενημέρωση υπάρχει. Αναφέρθηκε αυτός ο δημοσιογραφητής Αυτό εφαρμόζεται κάπως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα ήθελα να αλλάξει μέσω νομοθεσίας ευρωπαϊκής. Νομίζω ότι μόνοι μας μπορούμε να τα καταφέρουμε, δεν θα θέλαμε να αλλάξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκε και το θέμα αυτό ε, των ε, συμβάσεων μελλοντική απόδοσης. Εθελοντικά λειτουργήσε το σύστημα. Μα απογοητεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμίχθηκε σε αυτό. Η αγορά των futures δεν λειτουργεί εκτός αν υπάρχει κερδοσκοπία. Αυτό είναι ο στόχος της ύπαρξής τους. Πρέπει να υπάρχει κερδοσκοπία, ένα ποσοστό. Αν θέλετε να απαλλαγεί το διακύμαση των τιμών υπάρχει η κάθετη ολοκλήρωση. Αν θέλετε μπορείτε να το πετύχετε αυτό. Αν αυξηθεί η τιμή των ζωοτροφών αυτόματα μου δίνει υψηλότερη τιμή ε, στο ε, σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες απορρόφησης των κλειδονισμών. Υπάρχουν οι δυνατότητες αλλά α, χάνεις κάπως την ανεξαρτησία σου. Αυτά ήθελα να πω, ζητώ συγγνώμη αν τελικά μακρηγόρησα. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν να σας συγχαρώ για μερικά από τα συμπεράσματά σας, όπως για το συμπέρασμα που δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη για τη διαχείριση του κινδύνου. Ε, επίσης κάποιες προτάσεις που αφορούν τις αυτές εμπορικές πρακτικές είναι ενθαρρυντικές για το δίκαιο ανταγωνισμού πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπε ο κ. Σαμίρ και είπε ότι η απελευθέρωση των διεθνών αγορών θα είναι υποφελής ε, εφόσον ε, έχουμε ελεύθερο ανταγωνισμό μεταξύ χωρών ε, με αντίστοιχη οικονομική, αντίστοιχο οικονομικό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι κοινή λογική. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε στο παρελθόν να θέμε τις εμπορικές πρακτικές από τρίτες χώρες όπως ε, ανοίξαμε την αγορά ελαιολάδου μας στο τινησιακό ελαιόλαδο. Και μάλιστα ήταν προτάσεις που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που ζήμιωσαν το, το ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είχαμε λοιπόν τέτοια ανοίγματα αγοράς ε, για τα προϊόντα τρίτων χωρών που δεν ε, πληρούν αντίστοιχε υψηλέ προδιαγραφέ με του δικού μα γεωργού. Σκοπεύετε να κάμψετε ή να, ή να διακόψετε αυτή την πολιτική που είναι άδικη απέναντι στους ε, Ευρωπαίους Γεωργούς, υιοθετώντα κάπως πιο προστατευτικά για αυτούς μέτρα. Επίσης, ε, η αυτάρκεια επιστηστική του, της Ευρώπης ε, είναι στόχος ε, της ΚΑΠ. Παρ' όλα αυτά το σημείο, 2009, το σημείο 209 μιλά για μια ΚΑΠ που στο μέλλον θα πρέπει να αντιμετωπίσει κάποια έξω ευρωπαϊκά προβλήματα όπως είναι οι μεταναστευτικές ροές. Πιστεύετε ότι αυτός είναι ο ρόλος των γεωργών της κοινή γεωργικής πολιτικής να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της μεταναστευτικής κρίσης ή θα μετατρέψει την ΚΑΠ σε ένα εργαλείο στήριξη των μεταναστών. Νομίζω ότι τέτοιου είδους προτάσεις θα οδηγήσουν σε ένα τελείως δύσχριστο σύστημα που θα εκφύγει το ελέγχο. Μας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκίσεν, τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, της Ειδικής Ομάδας και στον Επίτροπο Χόγκαν και μετά και στους, στα μέλη τη ειδική ομάδα. Θα θέλω να απαντήσω σε συγκεκριμένε ερωτήσει στο μέλλον τη Επίτροπή Πρώτα λοιπόν θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο και στον κύριο Γκίσεν για να σχολιάσουν ή να απαντήσουν τι ερωτήσει των Ευρωβουλευτών. Δεν ξέρω ποιο θέλει πρώτο το λόγο. Ο κύριο Επίτροπο πρώτο, ο κύριος Χόγκαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλου για τα υποκοδομητικά του σχόλια. Στρέφομαι στου εμπειρογνώμονε των διαφόρων φορέων που εκπροσωπούνται. Θέλω να πω ότι τα στοιχεία που παρεσχέθησαν από τον πρόεδρο της ΚΟΠΑ δείχνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και γι' αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήσαμε αυτή την Task Force. Για να ανοιχνεύσει τα αίτια των προβλημάτων των γεωργών. Και τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μείωση του περιθωρίου του κόστους των συναλλαγών που βαρύνουν ε, το γεωργό και τι ρόλο παίζουν μεταποιητές και λιανοπολιτές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε την χρήση των οργανώσεων των παραγωγών. Και τονίζεται ιδιαίτερα αυτό. Τονίζεται η διαφάνεια της αγοράς και το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι οργανώσεις των παραγωγών. Το αναφέρουμε στις τάσεις. Εξετάζουμε θέματα ανταγωνισμού που περιγράφονται και ο Νταντέν αναφέρθηκε σε αυτά. 28 Φεβρουαρίου θα είμαι εδώ με την κύριε Βέστιγκερ την Επίτροπο, την υπεύθυνη περί ανταγωνισμού, για να δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε καλύτερα όσον αφορά τα προβλήματα της γεωργίας. Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στα διάφορα ζητήματα. Δεν θα απαντήσω ξεχωριστά στον κάθε, στον καθένα, αλλά θα αναφερθώ στην υποχρεωτική ενημέρωση όσον αφορά ΜΕΣΚ, μεγαλύτερη διαφάνεια, τυποποίηση των στοιχείων. Σε αυτά που είπατε θα αναφερθώ. Ποιότητα των στοιχείων. Το κόστος του κεφαλαίου. Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι αυτό τονίθηκε από πολλούς. Θα μπορούσε Προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αναπτύξει τα χρηματοδοτικά προϊόντα για τους γεωργούς. Βελτιώνεται η κατάσταση πρόσφατα, χάρη στις προσπάθειες. Αυτό είναι ευπρόσδεκτο. Έχουμε πολλά που μπορούμε να κάνουμε ακόμα. Ο καθηγητής Πένιγκ αναφέρθηκε στη διαχείριση του κινδύνου, διακύμανση των τιμών, κόστος κεφαλαίου. Αναφέρθηκε στη ΣΥΠΑ ότι χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία μας, ε, τη δική μας οι Αμερικανοί και δεν χρησιμοποιούμε εμείς αρκετά. Ίσως μπορούμε να το διερευνήσουμε αυτό. Τι ακριβώς σημαίνει. αν αυτό το χρόνο. Όσον αφορά τους συντονιστές, τους ευρωβουλευτές, όλοι δέχονται ότι τεπαιτείται δράση. Θέλουμε να το εξετάσουμε αυτό. Συνεργαζόμαστε στενά με την g και την Γενική Διεύθυνση, την υπεύθυνη του ανταγωνισμού επ' αυτών. Και στο κολέγιο των επιτρόπων θα συζητηθεί δεν θα εξετάσουμε μόνο τη γεωργία, θα πρέπει να καταλήξουν σε μια γενική πρόταση, η οποία θα βρίσκει και άλλους συμφώνους. Η δράση Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, υποστηρίζεται εδώ, με την εξαίρεση του κυρίου Άγνιου, του καλού μου φίλου, κάτι αναμενόμενο άλλωστε. Οι κλονισμοί ε, λόγω διακύμανσης των τιμών. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε βεβαιότητα το μέλλον. Βελτιώνεται όμως το συνέστημα σε τομείς που αντιμετώπισαν δυσκολίες ε, στο κάτω παρελθόν, στον τομέα του γάλακτος και του χειρίου. Θα ασκηθούν πιέσεις στους παραγωγούς βοήου. Ξέρουμε την εκλογική μας περιφέρεια ότι παράγοντες που σχετίζονται με τον Brexit θα επηρεάσουν τις τιμές. Θα πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση, να δούμε αν χρειάζεται παρέμβαση τα θέματα που εντοπίστηκαν στην έκθεση φαίνεται να τα υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό. Δεν άκουσα κάποιον να λέγει ότι υπάρχουν και άλλες προτάσεις που θέλετε να προσθέσετε στις συστάσεις. Αυτό δείχνει σαφώς ότι οι εμπειρογνώμονες έκαναν μια αρκετά καλή δουλειά, ετοίμασαν ε, ένα μενού ε, προτάσεων για μελλοντικές ε, νομοθετικές δράσεις. Είναι ανεξάρτητη έκθεση, το τονίζω αυτό. Ζητήσαμε από όλε τι γενικέ διευθύνσει του σώματος να εξετάσουν ανεξάρτητα τι και να δούμε τι συστάσεις μπορούμε να υποβάλουμε από το μενού που μας δίνει η έκθεση για να υποβάλουμε τις προτάσεις τους ε, γεωργού. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες ε, ερωτήσεις αλλά θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στο θέμα των προθεσμιακών αγορών, α, και αν μπορούν και οι συναδελφοί μου. Λοιπόν, πολύ σωστά νομίζω πως ε, είπε ο κ. Επιτροπός ότι με την έκθεση αυτή πλέον το μπαλάκι βρίσκεται στο γήπεδο της Κομισιόν αλλά και στο Κοινοβούλιο που βεβαίως ε, θα παρακολουθήσουμε την ε, εξέλιξη και πραγματικά θα θέλαμε να σας ενθαρρύνουμε να κάνετε περτερό επαφές. Να αφαιρθώ σε ένα ερώτημα για το ζήτημα των διακλαδικών αυτών οργανώσεων που υπάρχουν ειδικά στην Ισπανία ενώ υπάρχει ζήτημα και πρόβλημα θα έλεγα στη Γερμανία δεν έχουμε βρει ακόμα ένα επιτυχημένο τέτοιο παράδειγμα και θα ρίνουμε παρόλα αυτά να ε, ιδρυθούν αυτοί οι κλαδικοί ε, οργανώσει οργανώσεις, οι κλαδικές οργανώσεις των ε, αγροτών. Θετικό λοιπόν μήνυμα, αλλά βεβαίως το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει αυτά να γίνουν στο κάθε κράτος μέλος δεύτερον. Για το θέμα του ανταγωνισμού και των οργανώσεων αγροτών. Γεγονός είναι πως έχουμε δύο γενικές διευθύνσεις που είναι σε διάλογο γεωργίας και ανταγωνισμού. Εμείς μπορούμε να ενθαρρύνουμε, να σπάσουμε το 15% που ισχύει αυτή τη στιγμή ως όριο των παραγωγών και νομίζω πως εάν φτάσουμε σε ένα 33% της αγοράς ε, νομίζω πως ε, θα είναι κάτι το θετικό. Χρειάζεται λοιπόν αυτός ο διάλογος αλλά και να δημιουργηθεί μια ασφάλεια για να μπορούν και οι οργανώσεις να ξέρουν πώς θα κινηθούν στο μέλλον γιατί αλλιώς τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ ακριβά. Τέλος όπως είπαμε μπορούμε να δεχτούμε από τη είπα όσον αφορά τις, ε, τα συμβολία μελλοντική εκπλήρωσης αυτό το οποίο είπε ο κύριος ε, Χόσλινγκ, πράγματι οι τιμές και οι ποσότητες ε, πράγματι ε, είναι, έχουν μια σχέση τραμπάλας θα λέγαμε. Αλλά ποιος θα μειώσει τις ποσότητες, θα είναι ο μεμονωμένος αγρότης, θα είναι οι συνεταιρισμοί, θα είναι το κράτος. Εγώ θεωρώ πως θα πρέπει να το αφήσουμε αυτό στις αγορές που είναι πολύ πιο κοντά σε όλα αυτά από τον οποιονδήποτε πολιτικό γιατί ε, βλέπουμε το τι γίνεται και στις αγορές ε, του χοιρινού κρέατος που είχαν σχεδόν εξουθενωθεί πριν από ένα χρόνο και τώρα ε, βρίσκονται ξανά σε μεγάλη ανάκαμψη. Βεβαίω υπάρχει πράγματι ο κίνδυνος όπως αναφέρθηκε όσον αφορά την αλυσίδα αυτή της αξίας να βρεθούν σε θέση μισθωτού ή εξαρτώμενης εργασίας οι γεωργοί. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουν τι συμβάσεις οι γεωργοί για να αποκτήσουν περισσότερη δύναμη. Και τέλος κύριε Λουαζό, ε, δεν θέλουμε προστατευτισμό εμείς. Μηδέν. Θέλουμε άνοιχτες αγορές και δεν νομίζω πως ε, υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα εδώ πέρα. Πρέπει να αφήσουμε τις αγορές να λειτουργήσουν. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και στην εμπειρογνώμονα από, την ειδική ομάδα εργασία, αλλά παρακαλώ να είστε λακωνικοί. Κυρία Νίκο Ιουχάς. για τη διαφάνεια της αγοράς, καταρχήν για το κόστος. Ήδη καταβάλουμε υψηλό κόστος για τη συγκέντρωση των δεδομένων. Δεν θέλουμε να αυξήσουμε το κόστος. Θέλουμε να εναρμονίσουμε τη συγκέντρωση των δεδομένων και να διδαχθούμε από τις εμπειρίες μας για να έχουμε ένα είδος προτυποποίηση. Δεν θέλουμε αύξηση του κόστους, αλλά μια πιο ορθολογική δαπάνη των κονδυλίων. Επίσης, η συγκέντρωση των δεδομένων για τις τιμές εφαρμοζόταν για λόγους πολιτικής, για λόγους κοινής γεωρικής πολιτικής. Είναι όμως ε, από τις πιο σημαντικέ πληροφορίες που έχουν οι γεωργοί οι πληροφορίες για τις τιμές. Ε, και όχι μόνο για τους γεωργούς είναι σημαντικές είναι οι πληροφορίες για τις τιμές, αλλά και όλους τους κρίκους της ε, τροφικής αλυσίδας. Μάλιστα, με βάση μια έρευνα που έγινε, είναι μετά τον καιρό και αντίστοιχου σημαντικού παράγοντε, έρχεται τρίτο στη σειρά σε ό,τι αφορά τη σημασία το θέμα τη ενημέρωση, τη υποβολή στοιχείων για, το, για τι τιμέ. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια εναρμόνιση, πιο τυποποιημένη συγκέντρωση και διαφορετική εστίαση, να προσανατολισόμαστε περισσότερο στι ανάγκε του Γιώργου. Γι' αυτό κάναμε τι σχετικέ προτάσει. Για κανένα άλλο λόγο και όχι για την αύξηση κόστου σε καμία περίπτωση. Ο Επίτροπος ήθελε να απαντήσει και σε κάποιον άλλο ευρωβουλευτή που ξέχασε πριν. Συγγνώμη, ετέθησαν κάνα δύο ερωτήσεις. Το θέμα αυτό 30.000 τόνοι συμφωνήσαμε την, την Ισία για το ελαιόλαδο για δύο χρόνια. Στα μισά βρισκόμαστε τώρα. 19.900 τόνοι ήρθαν. Άρα η Τινήση δεν είναι πολύ ανταγωνιστική όσον αφορά τις αγωγές Ελαιόλαδο εν συγκρίση με τις χώρες Μεσογείου δεν υπήρχε αναστάτωση στην αγορά στη Βόρεια Ευρώπη. Για να βοηθήσουμε την Αφρική. Είναι στρατηγική απόφαση που ελήφθη προκαιρού. Πώς βοηθάμε την Αφρική. Για να μπορούν οι ίδιοι να, να παράγουν γεωργικά προϊόντα και να μειωθεί και η μετανάστευση στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει ξεκινήσει ένα σημαντικότατο πρόγραμμα με τη βοήθεια κρατών μελών για να δώσουμε χρήματα για να βοηθήσουμε τους γεωργούς. Οι περισσότερες είναι γυναίκες στην Αφρική, ούτω ώστε να καλλιεργούν καλύτερα, να έχουν σωστή τεχνολογία, να μπορούν να αποθηκεύουν τα προϊόντα τους, να καινοτομούν, για να μπορέσουν να θρέψουν τον αυξανόμενο πληθυσμό που αυξάνεται με πολύ γοργούς ρυθμούς στην Αφρική. Οι θα αντιμετωπίσουμε σοβαρότατο μεταναστευτικό πρόβλημα για άλλους λόγους, εκτός πολέμου στο μέλλον. Ήδη έχουμε προγράμματα αναπτύξεως υπαίθρου που δίνουν τη δυνατότητα να τα μεταβάλουν τα προγράμματα ανάπτυξης υπαίθρου ε, για να τα προσαρμόσει τοπικές ανάγκες ανάλογα με τη μετανάστευση κλπ. και τις διάφορες προτεραιότητες που έχει κάθε περιοχή και κάθε κάτω μέλος. Έχουν τη δυνατότητα κάτι μέλη να τροποποιούν το πρόγραμμα ε, της ανάπτυξης υπαίθρου για στέγαση ή για άλλες υπηρεσίες ούτω ώστε να προσαρμόζονται στι ανάγκε ε, και ανάλογα με την εισρωή των μεταναστών στη συγκεκριμένη περιοχή. Σα ευχαριστώ. Παίρναμε τώρα στα σχόλια των υπόλοιπων ε, ευρωβουλευτών. Ένα-ενάμιση λεπτό το πολύ. Αλλά όχι παραπάνω. Και αν έχουμε χρόνο θα ξαναδώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες. Ο κύριος Ντες, όπως είπα, ένα λεπτό, ενάμιση λεπτό το πολύ, όχι παραπάνω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και για τη δουλειά που έγινε εδώ πέρα. 12 χρόνια είμαι στο Κοινοβούλιο, 12 χρόνια ζητάω νομοθετικά μέτρα. Είναι καλό για τις ε, προθεσμίες πληρωμής, καλός είναι αυτός ο στόχος για τις 30 ημέρες ε, που θα πρέπει να ισχύσουν επί της αρχής για γάλα και κρέος. Ναι, καμία συμμετοχή λέτε στο κόστος επεξεργασίας και διάθεσης. Μα ε, τιμή, όταν λέμε τιμή εννοούμε την καθαρή τιμή, οτιδήποτε άλλο είναι αδιαφανές. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα απόλυτα προϊόντα, να μην αποθηκεύονται επίσης τα ευπαθή την τελευταία στιγμή. Και βεβαίως ε, θα πρέπει όλες οι εμπορικέ ε, πρακτικές στην Ευρώπη να είναι ξεκάθαρες ε, και για τους ε, πελάτες και για τους αγρότες. Και βεβαίως, όπως σας είπα, είχαμε το ανάλογο στα τσιγάρα, όπου ξέρουμε πόσοι είναι η τιμή και ο φόρος, κάτι ανάλογο θα πρέπει να υπάρχει και στο, στα τρόφιμα. Αυτό το περιθώριο κέρδους που αναφέρεται επίσης είναι τελείως αδιαφανές. Αυτά και θα υποβάλω και τις προτάσεις μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Επίτροπο. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω πρώτα την Task Force Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπόνηση της έκθεσης και τα συμπεράσματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις υπηρεσίες ε, με τις οποίες ε, είχα επαφές ε, κατά την εκπόνηση της έκθεσής μου για τα εργαλεία της κοινή γεωρικής πολιτικής προκειμένου να μειωθεί η αστάθεια των τιμών. Όπως ξέρετε, η έκθεσή μου εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία τον περασμένο Δεκέμβριο και χαίρομαι γιατί καταλήγουμε στα ίδια συμπεράσματα και στις δύο εκθέσεις, τη δική μου και τη δική σας. Γιατί ε, ε, προτείναμε τις ίδιες βελτιώσεις, να βελτιωθεί η θέση των παραγών στην ε, τροφική αλυσίδα, μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά, ένα καλύτερο εργαλείο για τη διαχείριση του κινδύνου, αποτελεσματική καταπολέμηση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών, αναθεώρηση του δικαίου ανταγωνισμού και ιδιαίτερα του άρθρου 40 του δικαίου ανταγωνισμού που θα πρέπει να γίνουν σεβαστά και η γεωργία να θεωρηθεί ως ξεχωριστός ιδιαίτερος τομέας ε, της οικονομίας. Ε, Επίση, σημαντικό είναι το θέμα της χρήσης των γραπτών συμβολέων για να επανισορροπήσουμε τη σχέση μεταξύ των διαφόρων κρίκων της τροφικής αλυσίδας. Επίσης, το μοντέλο των διακλαδικών ήδη επαγγελματικών οργανώσεων κατά τη γνώμη μου είναι ο καλύτερος τρόπος για να φτάσουμε σε μια ενισχυμένη χρήση των συμβάσεων. Παρόλο που είδαμε το θέμα λοιπόν από διαφορετικές σκοπιές, καταλήξαμε στα ίδια συμπεράσματα και στις ίδιες προτάσεις, κάτι που είναι πολύ θετικό για τη μελλοντική κοινή και ορική πολιτική. Τώρα περιμένουμε απτές προτάσεις από το Συμβούλιο, αλλά και από εσά κύριε Επίτροπε. Και δεσμεύομαι να λάβω μέρος ε, στο έργο που θα ξεκινήσει για το μέλλον της κοινή γεωρικής πολιτικής και ελπίζω τα συμπεράσματα και των διεκθέσεων να ληφθούν υπόψη στις μελλοντικέ σας προτάσεις. Ευχαριστώ. Η ομάδα εργασίας ε, έλαβε γνώση της έκθεσής σας και φαντάζομαι την εξέτασε, γιατί και εσείς πραγματευτήκατε το ίδιο και πολύ σημαντικό θέμα. Η κυρία Μαγκίνες τώρα. Ε, thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους όσους ε, μίλησαν. Ένα σχόλιο έχω. Δεν θα αναφερθώ σε αθέμητες εμπορικέ πρακτικές εκτενώς. Επίτροπε, φαίνεστε προσεκτικός όσον αφορά το πώς θέλετε να προχωρήσετε. Γιατί, διαρωτώ με γιατί. και ότι πρέπει να υποκριθούμε στη Γενική Διεύθυνση για τον Αγωνισμό και Εσωτερική Αγορά. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος σας βοηθά, διότι μιλάμε για βιώσιμη, βιώσιμο φοδιασμό σε τρόφιμα, οικονομικά βιώσιμα και περιβαλλοντικά βιώσιμο τομέα. Μπορείτε να το, να ξεκαθαρίσετε αυτό. Δεύτερον, κάτι που μας ενδιαφέρει. Οι προτάσει για το μελλοντικό τη κοινή αγροτική πολιτική, για το μέλλον τη κοινή αγροτική πολιτική. Πολλέ παράγραφοι 190 και 193 αναφέρονται λεπτομερώς αυτό Ποια είναι η άποψή σας επ' αυτού. Ποια είναι η άποψή σας για τις προτάσεις για τη μελλοντική ΚΑΠ. Οι συντάχτες διατείνονται ότι θα πρέπει να απομακρυνθούμε από άμεσες πληρωμές όσο έχουν και να έχουμε διαφοροποιημένα μέτρα στην αγορά. Σχόλιά σας θα θέλαμε. Το εγκρίνετε. Θέλετε να προσθέσετε κάτι σε αυτό που προτείνετε. Μάλιστα εσείς έχετε Είχατε, είχατε συντάξει και γνωμοδότηση για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και εκεί ε, παρουσιάζεται εκτεταμένα τις απόψεις. Η κυρία Κόστιγκερ. Ευχαριστώ. Νομίζω όλοι αναμέναμε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και να ευχαριστήσω τον κύριο Γκίσεν και έχει δίκιο. Όλοι θα ευχόμασταν να δρουν οι αγορές, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι συχνά την δύναμη των μονοπωλίων και έχουμε εκατομμύρια αγρότες που πλέον δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν εισόδημα από τις τιμές της αγοράς. Το πρόβλημα το οποίο βλέπουμε παντού από το βορρά στο νότο, την Ανατολή ω τη Δύση είναι πως οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν τόσο μεγάλη πίεση ώστε πλέον απειλείται η ύπαρξή τους, οι επιδοτήσεις γίνονται όλο και μικρότερες, οι απαιτήσει όλο και μεγαλύτερες, ε, ευζοία των ζώων, περιβάλλον και τα λοιπά και πάρα πολλά από αυτά νομίζω φαίνονται στην ανισορροπία που υπάρχει και νομίζω είναι σαφές ε, και άρα το ερώτημα προς εσάς ε, κύριε Επίτροπε είναι μήπως υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για ε, μέτρα, εφαρμογή, γιατί ακούμε για εθελοντικά μέτρα, επαναλαμβάνεστε συνεχώς ε, εθελοντικά, εθελοντικά, δεκάδες φορές Θα έχουμε πει. Επίσης ρητά στο πρόγραμμα εργασίας κομισιών αναφέρατε πως θα πρέπει να γίνουν κάποια μέτρα προς αυτή η κατεύθυνση όσον αφορά τη διαφάνεια της αγοράς, τις ε, αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ, τι πρακτικέ των συμβάσεων και οπωσδήποτε το δίκαιο του ανταγωνισμού. Ε, θα μπορούμε να περιμένουμε νομοθετικές ε, πρωτοβουλίε φέτο. Ευχαριστώ, Αράντς Καρσία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχηθώ στον Επίτροπο και σε όλους σας ευτυχισμένος ο καινούριο χρόνος, ευτυχισμένο το 2017, γιατί οι προτάσεις που θα υποβάλλετε για την ΚΑΠ μετά το 2018 θα αρχίσουν να διαμορφώνονται στο μυαλό σας ήδη από φέτος, από το 2017. Γι' αυτό σας εύχομαι καλή τύχη και καλή χρονιά για όλους μας ε, και για τους ε, γεωργούς που περιμένουμε πώς και πώς προτάσεις. Εγώ θα μιλήσω για τα συστήματα διαχείρισης ε, κινδύνων που στηρίζονται σε συστήματα ασφαλίσεων και αμοιβαιοποίησης. Θα πρέπει να συμπληρώνουν και να μην αντικαθιστούν το πρόγραμμα αμέσων ενισχύσεων που έχουμε σήμερα. Και τα συστήματα αυτά ασφάλισης και αμοιβαία ασφάλισης θα πρέπει να είναι συμβατά με τα εθνικά συστήματα ασφάλισης για να μην διαταραχθούν ε, πράγματα που λειτουργούν ήδη καλά. Ποια είναι η γνώμη σας κύριε Επίτροπε. Επίσης ε, το παρατηρητήριο διαχείριση των τιμών, αλλάζω τώρα θέμα, που έχουμε για το χείριο κρέας ή για το γάλα θα μπορούσε να αποτελέσουν υπόδειγμα και για άλλους τομείς όπως και τα ποροκυπευτικά, που όπως γνωρίζετε είναι ένας κλάδος που αντιμετωπίζει μια πολύ λεπτή κατάσταση λόγω των ε, τιμών, λόγω των επιθέσεων που έχει υποστεί, λόγω της μεγάλης ανασφάλειας που επικρατεί στα απορροκυπευτικά, αλλά και λόγω των πιέσεων και των εξωτερικών παραγόντων. Για παράδειγμα, επιζωτίες που, που εισάγονται από τρίτες χώρες και που πλήττουν τον κλάδο των προκυπευτικών. Θα έχουμε προτάσει ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροφική Ελισίδα, όπω αυτές που έχουμε στην Ισπανία, με κυρώσει ε, ώστε να ε, χαλιναγωγήσουμε και να τιμωρήσουμε τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Θα υποβληθούν σχετικές προτάσεις από την Επιτροπή, κύριε Επίτροπε, ο κύριε Ράιερ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε και στα μέλη της να δώσω συγχαρητήρια. Έχω δύο ερωτήσεις ε, θα ήθελα οι επιχειρήσει μας και οι αγρότε μας να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια του Ταμείου Γιούνκερ, το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έχουμε 600-700 ε, δισεκατομμύρια στο σχέδιο αυτό, τα οποία δεν μπορούν να πάνε στους ε, γεωργούς με κανέναν τρόπο. Και μετά μιλάμε, δεν ξέρω, τι μπορεί να γίνει και για την Βασιλεία 3 και για το επαρκές ε, κεφάλαιο. Μετά. Όταν μιλάμε για μια αλυσίδα παραγωγής, ε, κοιτάξτε, ε, δεν έχουν πρόβλημα στην Ολλανδία με αυτό, αλλά λένε ότι θα θέλουν να διατηρήσουν την δύναμη οι αγρότες. Αυτός είναι ο, ο στόχος. Μπορείτε να μου υποσχεθείτε κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και κύριος που ήσταν σύντομοι. Ο κύριος Μπούντα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχηθώ καλή χρονιά και να εκφράσω τη χαρά μου για την προσπάθειά μας να ενισχύσουμε τη θέση των γεωργών παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού. Χαιρετίζω και τα συμπεράσματα της έκθεσης και ελπίζω να υιοθετηθεί και ένα χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των πολυχρήσιμων αυτών συστάσεων. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε κάποια στοιχεία της ρουμανικής πραγματικότητας. Στη Ρουμανία εγκρίναμε νομοθεσία για να ενισχύσουμε την θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ζητήσαμε από τα, τις, τα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, να αγοράζουν ε, τοπικά τα προϊόντα τους, όσο πιο κοντά γίνεται την τοποθεσία τους. Κάτι που ε, δημιουργεί ωφέλη και για τον παραγωγό και για τον καταναλωτή. Παρ' όλα αυτά, οι μεγάλες αλυσίδες διανομής δεν αντέδρασαν καλά όπως περιμέναμε. Μάλιστα, ο Επίτροπος μας απείλησε να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εις βάρος μας. Κάτι που μας εξέπληξε, γιατί και άλλα κράτη-μέλη έχουν λάβει παρόμοια μέτρα. Όταν δραστηριοποιούνται τα κράτη για να ενισχύσουν τη θέση των γεωργών θέλετε να τα τιμωρήσετε. Δεν είναι παράδοξο αυτό. Θα πρέπει να είμαστε έντιμοι και ειλικρινεί όταν λέμε ότι θέλουμε να ενισχύσουμε τη θέση του γεωργού στην αλυσίδα ανεφοδιασμού και δεν θα πρέπει να περιοριστούμε σε ωραία λόγια και να περιεχομένου. Ευχαριστώ. κύριο Ντόρφμαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η δουλειά της Task Force είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και τώρα θα πρέπει να βρεθεί ένα σχέδιο εφαρμογής, ε, το οποίο βεβαίω δεν είναι δική τους δουλειά, αλλά θα πρέπει να μην καταλήξει πάλι και αυτή η πρόταση σε ένα σιρτάρι. Έχω πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Αναφέρθηκαν ε, πολλές φορές οι κανόνες του ανταγωνισμού. Σήμερα στην κοινή γεωρική πολιτική έχουμε πολλές ε, περιπτώσεις όπου προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ε, προσφορά. Θα αναφέρω δύο πράγματα. Την αγορά οπορο Ο προσπαθούμε να δούμε πώς θα συνενωθεί η παραγωγή πολλών εκμεταλλεύσεων και δεύτερο αυτό που κάναμε πριν από λίγα χρόνια το ζήτημα της ε, παραγωγής ε, του ε, γάλακτος, όπως προσπαθήσαμε να το συνδέσουμε οπωσδήποτε με το ζήτημα και της ε, ονομασίας προέλευσης. Μήπω θα μπορούσαν να επεκταθούν τέτοια συστήματα και σε άλλα προϊόντα. Νομίζω πως είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Κυρία Χόιμπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. να αναφέρατε πως ε, θέλετε να αφήσετε την ρύθμιση στις αγορές, αλλά η κρίση νομίζω κατέδειξε ε, πως ε, τελικά αυτά τα πληρώνουν πάντα οι ίδιοι, όπως παραδείγματος χάρη η παραγωγή του γάλακτος. Νομίζουμε πως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ήταν πάρα πολύ έντονες, πάρα πολλοί γεωργοί σταμάτησαν την ε, παραγωγή, οπότε το να τα αφήσουμε όλα στις αγορές είναι μια κακή ε, απόφαση. Μιλήσατε επίσης για τα θέματα των συμβάσεων, αλλά βλέπουμε στην Γαλλία όπου εργάζονται με συμβάσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν καλύφθηκε το κόστος των αγροτών. Οπότε αν ε, δεν περιλαμβάνεται το κόστος ε, της, ε, της διατήρησης της ζωή των αγροτών, τότε δεν έχουν καμία αξία αυτές οι συμβάσεις. Και πώς θα μπορέσουμε οι αγρότες στην Ευρώπη να ανταγωνιστούν όταν υπάρχουν περιοχές στην Ευρώπη όπου δεν υπάρχουν ακόμα ε, δεν υπάρχουν, παραδείγματος χάρη ο κάθε αγρότης ε, έχει μόνο έναν αγοραστή για το προϊόν του. Δεν υπάρχει πουθενά δεύτερος και δεν υπάρχει δυνατότητα να συνεταιριστεί με κάποιον άλλον. Πώς θα μπορέσουν έτσι να... Πώς μιλάμε για δίκαιο ανταγωνισμό και να κοιτάνε στα μάτια τους αγοραστές τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Καλή χρονιά και από μένα. Νομίζω πως είναι το σημαντικότερο θέμα αυτό για την Γεωργία συνολικά. Προσφάτως ήμουν σε μια διάσκεψη στην Αφρική όπου το θέμα ήταν το εμπόριο είναι πόλεμος. Ε, όταν περιγράφεται το εμπόριο ως πόλεμος αντιλαμβάνεται πως τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θα πρέπει τουλάχιστον λοιπόν να έχουν και οι εμπορικοί εταίροι μας ε, τα ίδια όπλα. Και βεβαίως εδώ πέρα ακριβώς ε, η παραγωγή και η ενδιάμεση δεν έχουν τα ίδια όπλα. Γιατί μιλάτε από τη μία η κατάχρηση της ε, αγοράς και από την άλλη για διαχείριση του κινδύνου. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα διαχωρίσουμε ξεκάθαρα. Η διαχείριση του κινδύνου, ε, κάτι το οποίο είναι πολιτικά επιθυμητό, δεν έχει στόχο να αντισταθμίσει τις αποτυχίες της αγοράς. Έχει στόχο να αντισταθμίσει, παραδείγματο χάρη, τι καιρικέ καταστροφέ, ή ζητήματα πολιτικά όπω συζητήματα ζητηματα πολιτικα οπω η κατασταση με τη Ρωσία, αλλά όχι την ανισορροπία τη αγορά. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μα πείτε κάτι από αυτό. Υπάρχει ο ένα τομέα που είναι ότι πρέπει να λειτουργεί η αγορά και οι δύο συμμετέχοντε σε μια αγορά να έχουν αν θέλετε τα ίδια όπλα και βεβαίω να, να μπορούμε να αντισταθμίσουμε του κινδύνου, αλλά να μην περιγράφουμε ω κίνδυνο τις ελλείψεις της ε, αγοράς. Θα ήθελα δύο λόγια, γιατί συχνά τα μπλέκουμε αυτά τα πράγματα. Ποιο δημιούργησε αυτή τη σύγχυση. Ο κ. Φλάνναγκαν. Νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά των παραγωγών. εμεί παράγουμε. Αυτό πρέπει να ρωτήσουμε το εξής. Σαμένο τη GUNGL Τη αριστερή ομάδα αισθάνομαι παράξενο που θέτω την ερώτηση. Γιατί δεν μπορούν να έχουν χρηματοδο... πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι γεωργοί καταρχάς. Οι γεωργοί θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση αν ήταν ε, κερδοφόροι. Και εκείνοι δεν θα είχαν, ε, που έχουν τα χρήματα δεν είχαν πρόβλημα να διαδοτήσουν. Αντί να δημιουργούμε τεχνητέ καταστάσει όπου οι γεωργοί μπορούν να χρηματοδοτηθούν, σε περιπτώσει όπου δεν έχουν κέρδο, θα πρέπει να κάνουμε κάτι για το γεγονό ότι δεν έχουν κέρδο και να μιλήσουμε για όπλα. Είναι απλώς ποια είναι τα όπλα, πρέπει να είναι τα όπλα. Οι παραγωγοί θα πρέπει να παίζουν με ισότιμες συνθήκες, με τα εργοστάσια και εναντί των ε, υπεραγορών. Αυτή είναι η απλή απάντηση. Η ερώτηση τώρα. Υπάρχει προθυμία να το κάνουμε αυτό. Υπάρχει προθυμία να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Ή δεμή τότε το σημαντικότερο κομμάτι της αλυσίδας θα φύγει. Τα καλά μαντάτα, όπως ανέφερα και το επαναλαμβάνω, τα καλά, πολύ καλά μαντάτα ποια είναι. Ότι υπάρχουν χρήματα που βγαίνουν από τα τρόφιμα. Τα κακά μαντάτα δεν πάνε τα χρήματα στους σωστούς ανθρώπους. Δουλειά μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα πηγαίνουν στους σωστούς ανθρώπους. Υπάρχουν τα χρήματα. Θα πρέπει να ξαναπάνε στα χέρια της πρωτογενούς παραγωγής, του παραγωγού. Ο Στάκουλα. Ευχαριστώ. Ε, η προσπάθεια της βιομηχανίας να προασπίσει τα δικαιώματα των ε, λιανεμπόρων ε, δημιουργεί φοβερές ανησυχίες. Ε, γι' αυτό έχουμε άυξη των τιμών σε πολλά προϊόντα στα μαγαζιά λόγω των ιδιωτικών ε, ετικετών, των, των προϊόντων του σούπερ μάρκετ. Είχατε καθόλου συζήτηση στην ομάδα εργασία για τον κίνδυνο που δημιουργούν αυτές οι δυτικέ ετικέτες ε, στον κλάδο, γιατί η παραγωγή, οι συνεταιρισμοί ε, και ο κλάδος γενικός ε, θα υποστεί μεγάλες ζημίες αν επιτρέψουμε ελεύθερα στους σούπερ μάρκετ να μπορεύουν τα δικά τους προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές. Επίσης θέλουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αλυσίδα εφοδιασμού. Έχετε κάποιες προτάσεις για τον οικονομικό αντίκτυπο που είχαν οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές ε, στον αγροτοεπιστηστικό κλάδο. Γιατί πού είχαμε τις ε, μεγαλύτερες βελτιώσεις ε, με πανευρωπαϊκές ε, διατάξεις και τι οικονομικές συνέπειες ε, θα είχαμε σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης από μια τέτοια ρύθμιση. Ναι, κύριε Γκίσεν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την έκθεση της ε, Task Force. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι κάνατε συγκεκριμένες προτάσεις. Ατομική ευθύνη και διαχείριση κινδύνου για μένα δεν είναι αντίφαση. Ναι, έχει δίκιο η κυρία Νόχελ βεβαίω. η αποτυχία τη αγοράς δεν μπορεί να καλυφθεί από την διαχείριση κινδύνου. Το θέμα βεβαίως είναι μετά από πού θα βρούμε τα λεφτά. Εγώ είμαι κατά του να αφαιρεθούν χρήματα από τον πρώτο πυλώνα. Επίσης οι αγορές ε, ε, οι αγορές ε, μελλοντικής εκπλήρωση χρησιμοποιούνται μόνο από τους γαλακτοπαραγωγούς ε, που υπάρχουν πραγματικά διαπραγματεύσεις και καθορισμός ποσοτήτων σε συγκεκριμένο χρόνο και όταν ε, βεβαίως φύγαμε από τις ποσοστώσεις στον τομέα αυτών μάθαμε πολλά πράγματα για το πώς πρέπει να λειτουργήσουν καλύτερα οι αγορές και βέβαια χρειάζονται και μια σιγουριά οι ε, οικογένειες των αγροτών μας ε, και θα πρέπει να ενισχύσουμε την Ήπεθρο για να διατηρηθούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα να παραμείνουν στην Ήπεθρο και νομίζω πόσο καλό θα είναι να υιοθετήσει αυτές τις ε, προτάσεις στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ για την έκθεση αυτή της ομάδας κρούσης. Έχω μία παράκληση και δύο ερωτήσεις. Η παράκληση είναι προς εσάς ε, κύριε Επιτροπέ. Τι μπορούμε να περιμένουμε ως νομοθετική πρωτοβουλία. Ακούσαμε μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και μπρος. Μιλήσατε για υποδείγματα συμβάσεων, ε, για τον καθορισμό των τιμών, για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, αλλά πρέπει να δούμε και κάποια νομοθετική πρωτοβουλία. Και βεβαίω να συνοηθούμε και με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αν χρειάζεται βοήθεια οπωσδήποτε θα σας βοηθήσουμε και εμείς ε, Κατόπιν έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, η παρέμβαση. Για μένα είναι πάρα πολύ αργή η μηχανισμοί παρέμβασης που έχουμε σήμερα. Έχετε κάποια ιδέα για το πώς μπορούμε να παρεμβαίνουμε πιο γρήγορα. Γιατί τώρα από ό,τι φαίνεται το περιλαμβάνουν οι αγορές στις τιμές τους ότι θα υπάρξει κάποια παρέμβαση. Και τέλος, Βεβαίω υπάρχουν και τα λεγόμενα συστήματα πιστοποίηση ε, ε, που επιβάλλουν ε, διάφορα πράγματα στους αγρότες όταν μιλάμε δηλαδή για τις διαφορές αλυσίδες που θέλουν να αγοράζουν τα γεωργικά προϊόντα και που φτάνουν στα όρια της στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να γίνει εκεί πέρα. σα ευχαριστώ. Η κυρία Αγγιλέρα για ένα λεπτό. Δεν είχα σκοπό να ξαναζητήσω το λόγο, αλλά πρέπει να απαντήσω σε κάτι που είπε ο Επίτροπος Χόγκαν για το την Ισιακό Ελαιόλαδο, για να μην μείνει αναπάντητο το σχόλιο σας. Είπατε ότι στη τελική ανάλυση δεν κατακλειστήκαμε από την νησιακό ελαιόλαδο στην ευρωπαϊκή αγορά. Ε, μπήκαν πολύ χαμηλότερες ποσότητες από αυτές που αρχικά είχαν προβλεφθεί. Οπότε είπατε για τον Νότο δεν υπήρξε πρόβλημα ε, για τους παραγωγού παραγωγούς της Νότιας Ευρώπης. Ε, μιλήστε και για τα μέτρα για την Αφρική. Συμφωνώ με αυτά, αλλά διαφωνώ με αυτό που είπατε ε, και θα ήθελα να το επισημάνω εδώ. Οι Ευρωπαίοι γεωργοί και όσοι πασχίζουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση της γεωργίας στην Ευρώπη δεν είμαστε κατά των συμφωνιών με τρίτες χώρες ή με αφρικανικές χώρες γενικώ. Πάντως, όταν δεν τηρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις, όταν δεν πληρούνται οι ίδιοι όροι α, στις τρίτες χώρες με τις α, που ισχύουν εδώ, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για θεμητό ανταγωνισμό, γιατί τα στοιχεία, ε, τα κριτήρια της ασφάλειας, της υγιεινής, ε, τα περιβαλλοντικά κριτήρια είναι πολύ αυστηρά στην Ευρώπη και δεν μπορούμε να έχουμε πιο χαλαρές διατάξεις για τα θέματα αυτά σε τρίτες χώρες και να μιλούμε ε, για ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ ευρωπαϊκών και εξωευρωπαϊκών προϊόντων. Δεν μας προβληματίζουν ούτε το ελαιόλαδο της Τινησίας, ούτε τα πορτοκάλια της Νοτιοαφρικής. Αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι παράγονται σε διαφορετικές συνθήκες. Ούτε οι, ε, ε, οι Ευρωπαίοι Γεωργοί δεν θέλουν να βοηθήσουν την Αφρική ή την Αφρικανική Γεωργία. Απλώ είμαστε κατά το θέμα του ανταγωνισμού, γιατί τέτοιο de facto ισχύει, και οι συνθήκε είναι διαφορετικέ. Η κυρία Πετήρ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Οι συστάσεις της Ειδικής Ομάδας Εργασίας με τα συμπεράσματα της Επιτροπής και του Συμβουλίου, αλλά και με τις δικές μας προτάσεις, θα ενισχύσουν τις ε, γνώσεις που έχουμε για τον κλάδο και θα ενισχύσουν και τη θέση των παραγωγών. Γιατί αν δεν ενδιαφερθούμε εμείς για τους ε, γεωργούς, ποιος θα ενδιαφερθεί. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους γεωργούς στο έλεος της αγοράς η γεωργία εξασφαλίζει ε, τα τρόφιμα και ο αναφαντασμό σε τρόφιμα είναι ζωτική σημασία θέμα για κάθε χώρα. Οι γεωργοί δεν είναι μόνο επιχειρηματίες, έχουν σημαντικό ρόλο γιατί διαφυλάσσουν και την ε, εθνική ταυτότητα της κάθε χώρας. Επίσης, ε, θα πρέπει να τηρήσουμε την ισχύουσα νομοθεσία γιατί υπάρχει οδηγία που προβλέπει την πληρωμή μέσα σε 30 μέρες και είδαμε από τις συζητήσεις ότι δεν ε, εφαρμόζεται επαρκώς αυτή η οδηγία. Υπάρχει διαφορά επίσης στην ποιότητα των προϊόντων, είτε γεωργικών είτε άλλων, μεταξύ ε, των παλιών και των νέων χωρών μελών. Πραγματικά για τέτοια προϊόντα υπάρχουν διαφορετικές ποιότητες ε, και αυτό είναι διακριτική μεταχείριση και θα πρέπει να εφαρμοστούν οι ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, το θέμα των των εμπορικών πρακτικών. Βλέπουμε πώς αντιμετωπίζουν τα σούπερ μάρκετ ε, τους γεωργούς. Ε, γίνονται καταγγελίες ε, ή ακυρώσεις ε, συμφωνιών τελευταία στιγμή, αναδρομικές ε, τροποποίησεις. Αυτό είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει να χαλιναγωγήσουμε, να πατάξουμε τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, θα ήθελα να θαρρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιηθεί σχετική νομοθεσία για τους νέους γεωργούς, γιατί παραπονιούνται οι νέοι γεωργοί, όχι μόνο από την Κροατία, αλλά και από άλλες χώρες μέλη, ότι η σχετική νομοθεσία δεν τους επιτρέπει να ε, χρησιμοποιήσουν κονδύλια από, τα, από το κεφάλαιο της γεωργικής ανάπτυξης, κάτι που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μείνουν οι νέοι στην Ήπεθρο. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των αγορητών και θα δώσω τώρα το λόγο στους καλεσμένους, αλλά πρώτα, όπως πρότεινε και η κυρία Μαγκίνε, στον εκπρόσωπο της Ιρλανδικής Ένωσης Γεωργών. Και αυτό θα ακούσουμε. Τον κύριο Τζο Χίλι, παρακαλώ. Oh, Please Thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ καλωσορίζω την ε, αφοσίωση του Επιτρόπου του κ. Χόγκαν που θέλει να υλοποιήσει τα όσα αναφέρει η έκθεση και ταχύτερα δυνατόν Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δώσει δικό χάρτη η έκθεση περιέχει σημαντικές συστάσεις για αύξηση τη διαφάνεια στις τιμές και ανεξάρτητη εφαρμογή των μέτρων για ενισχυθεί θέση των γεωργών στην αλυσίδα των τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει υποβολή τιμών για γαλακτοκομικά, προκυπευτικά, κρέας και ε, λαχανικά για να μπορούμε να βλέπουμε ξεκάθαρα ποια είναι η διαμόρφωση των τιμών και τα κέρδη. Υποστηρίζω τις συστάσεις για αποτελεσματική και ανεξάρτητη επιβολή των μέτρων και του κανονισμού για την τιμή λιανικής και να προταθούν νέοι κανόνες σε, ευρωπαϊκό ε, επίπεδο για την προστασία από αθέμητες πρακτικές. Έχουμε νομοθεσία στην Ιρλανδία που θεσπίστηκε πέρσι. Ελήψη απαγόρευσης πωλήσεως κάτω του κόστους ε, οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα. Θα πρέπει οι προμηθευτές να έχουν την πεποίθηση ότι οι καταγγελίες θα διερευνώνται, ότι θα συμμορφώνονται οι αρμόδιοι με τον νόμο και θα επιβάλλονται οι κυρώσει όταν διαπιστώνονται καταχρήσει. Εν κατακλείδη, Πρόεδρε, εμεί οι Γεωργοί χρειαζόμαστε συστάσει εκθέσεω. Θέλουμε να εφαρμοστούν τι συστάσει, ώστε να επικρατήσει δικαιοσύνη σε λυσίδα των τροφίμων και να υπάρχει και σωστό επιμερισμό των κερδών. 21 εκατομμύρια Γεωργοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράγουν τρόφιμα για 500 εκατομμύρια καταναλωτέ, αλλά απολούν μόνο σε 110 ε, αγοραστικούς φορείς. Είναι πολύ συγκεντρωμένος ο τομέας της αγοράς των τροφίμων. Εκείνοι που αγοράζουν τα τρόφιμα είναι λίγοι, οι φορείς. Σας ευχαριστώ. Από τη Eurocommerce ε, ζήτησε το λόγο ο κύριος ε, Κριστήλεχρε. Κυρία μάλλον, είναι παρούσα η πρόσωπος της Eurocommerce, η πρόεδρος γιατί μας είχαν ενημερώσει για τη συμμετοχή του εκπροσώπου της Eurocommerce. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκπροσωπώ τη Eurocommerce στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους λεωπολιτές ε, και τους πολιτές χοντρική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχαρητήρια την οργάνωση Ακροάσεως. Άκρος ενδιαφέρουσα υπήρξα. Ακούσαμε πολλά σωστά σημεία στη συζήτηση. Συγχαρητήρια. Επίσης για τις συστάσεις της ομάδας ειδική για το θέμα των τιμών του αγροτροφομικού τομέα συμφωνούν πολλές συστάσεις εκτός από ένα κεφάλαιο το κεφάλαιο για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Δεν κατανοούμε γιατί εστιάζεται το κείμενο στις εμπορικές πρακτικές και γιατί θα πρέπει τα προβλήματα να αντιμετωπίσουν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμφωνούμε των γενικών θεμάτων όσον αφορά τις συστάσεις της ειδικής ομάδας. Θα πρέπει οι γεωργοί να έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη. Πρέπει να μπορούν να παράγουν με καλύτερα με καλύτερε διαγραφέ ποιοτικέ. Θα πρέπει να υπάρχει πιο σωστή διαχείριση των κινδύνων. Θα πρέπει να του βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Συμφωνούμε σε κάποιο βαθμό ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά. Πρέπει να εξηγήσουμε τι σημαίνει όσον αφορά την παραγωγή στην εκμετάλλευση και τη διαμόρφωση της τιμής λιανικής, απογοητευόμεθα από τα στοιχεία που ακούσαμε, είναι σφαλμένα όσον αφορά την κατανομή της προστιθέμενης αξίας. Χρειάζεται συζήτηση πράγματι. Πρέπει να δούμε από πού προέρχεται η προστιθέμενη αξία, πώς συνεργάζονται οι διάφοροι τομείς και πώς μπορούν να συνεργαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη του καταναλωτού για ποιοτικά προϊόντα σε προσιτές τιμές. Αυτό χρειάζονται οι λιανόπολιτές, να δίνουν στους καταναλωτές αυτό που επιθυμούν στα καταστήματά τους. Τώρα η ρύθμιση των εμπορικών πρακτικών δεν θα προστατεύσει τους γεωργούς από ιανδήποτε κρίση, ούτε θα τους προσφέρει μια καλύτερη τιμή. Οι πρακτικές που εντοπίζονται στην έκθεση δημιουργούν μεγάλες ανησυχίες. Αντικατοπτρίζουν γενικά τις σχέσεις των λιανοπολιτών με τους μεγάλους μεταποιητές και όχι με τους γεωργούς. Οι εμπορικές πρακτικές καλύπτονται σημαντικά από εθνική νομοθεσία όσον αφορά τον ορισμό τους, και όσον αφορά το πλαίσιο για την επιβολή των καταλήλων μέτρων. Επειδή οι λιανοπολιτές πολύ συχνά κινούνται σε εθνικό επίπεδο, το να φέρετε το 80% εδώ σαν στοιχείο, δεν είναι σωστό. Δεν υπάρχει συνοριακό πρόβλημα, άρα δεν μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ό,τι σε εθνικό. Άρα μια, ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν θα εξασφαλίζει ισότιμους όρους τα κράτη-μέλη και το τρόπος θα μπορούν να, να ομαδοποιούνται και να δημιουργούν προβλήματα όσον αφορά τον κατακαιρματισμό της αγοράς. Θα πρέπει η συζήτηση να εστιάζεται επί των βασικών θεμάτων. Υποστηρίζουμε τη δημιουργία σωστού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο. Σε διακλαδικό επίπεδο οι διακλαδικές οργανώσεις είναι ένα σημαντικότατο βήμα όταν υπάρχουν, αλλά μπορούν να υπάρξουν και άλλες προσεγγίσεις. Ο διάλογος για καλύτερη εξισορρόπηση ζήτηση και παραγωγής όσον αφορά την ποσότητα, την ποιότητα και την υποστήριξη για την καινοτομία είναι μια σωστή προσέγγιση. Ε, ήταν σημαντικό να ακούσουμε και εσάς, την εκπρόσωπο δηλαδή των εμπόρων, γιατί πιστεύω ότι, θέλουν, ότι χρειαζόμαστε το διάλογο μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της αλυσίδας. Δεν θέλουμε να μιλάμε μόνο μεταξύ μας. Θέλουμε πραγματικό διάλογο και εταιρικέ σχέσεις ε, μεταξύ των διαφόρων κρίκων αυτής της αλυσίδας της τροφικής. Και θα σας παρακαλούσα να μου στείλετε και γραπτό στα σχόλιά σας. Γιατί αυτό είναι ο στόχος μας για το ζητούμενο. Να έχουμε διάλογο επικοδομητικό μεταξύ μας. Γι' αυτό και ζητούμε και γραπτό στο κείμενο για να ληφθείτε όντω υπόψη. Και δεν είναι θέμα ποιο θα πείσει τον άλλο για τα επιχειρηματά του, θέμα είναι να γίνει διάλογο. Θα ακούσουμε λοιπόν του εμπειρογνώμονε μα. Ζήτησε το λόγο πάλι και ο κύριος Ντε. Ένα λεπτό όμω και μετά οι καλεσμένοι μας για δύο λεπτά ο καθένα. Ο κύριο Ντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πως το Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο και την Κομισιόν παρενέβησαν στις ε, αγορές γιατί οι εταιρείε δεν ήταν διατεθειμένες να καταργήσουν τα τέλη περιαγωγής. Πριν από χρόνια λοιπόν ξεκινήσαμε αυτή η διαδικασία και ε, μιλάμε για μεγάλη παρέμβαση στην αγορά. Το αναφέρω για να ενθαρρύνω τον Επίτροπο να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για να επιλύσει αυτή την δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί όσον αφορά ακριβώς την εμπορική δύναμη που έχουν απέναντί τους οι μεγάλες επιχειρήσεις. Πρέπει να ληφθεί μια νομοθετική πρωτοβουλία όπως κάναμε και για την περιαγωγή των κινητών τηλεφώνων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για το μεγάλο ενδιαφέρον, για τη συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση, λέει και ο Μέριλτ. Ευχαριστώ για όλα τα θετικά σχόλια που ακούστηκαν για τους Ευρωπαίους Γεωργούς. Χάρηκα που τα άκουσα αυτά. Αυτό μου δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την προστασία των Ευρωπαίων Γεωργών. Να υπογραμμίσω εκ νέου ότι είναι σημαντικό σε κάποια ζητήματα να κινούμεθα μέσω νομοθεσίας, αλλά πρέπει να κάνουμε και ό,τι μπορούμε, όπως προανέφερα, για να ανθαρρύνουμε τους γεωργούς να είναι πιο συνεργάσιμοι, να είναι πιο πρόθυμοι να συγχωνεύσουν κάποιους λειτουργούντες συνεταιρισμούς. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους διευκολύνουμε για να αρθούν τα εμπόδια από το δρόμο τους Κάποιοι κανονισμοί τους δημιουργούν προβλήματα, το ξέρουμε, αλλά υπάρχει και θέμα κατανόησης. Πρέπει να κατανοήσουν ότι πρέπει να συνεργάζονται οι γεωργοί. Και εμείς θα κάνουμε αυτό που μας αρμόζει. Χρειαζόμαστε όμως και υποστήριξη και από το πολιτικό σύστημα. Γι αυτό. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Πρόεδρε, να θέλω να επαναλάβω την έντονη αυτή συζήτηση. Νομίζω πως είναι καλές οι προτάσεις της ε, ομάδας κρούσης και καλό είναι να μην υπάρξουν νέα εμπόδια ε, για να ενεργοποιηθεί εδώ πέρα το ευρωπαϊκό και τα εθνικά επίπεδα. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε περισσότερη διαφάνεια για τις τιμές και βεβαίως για τις διαδικασίες παραγωγής. Μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, έτσι και βεβαίω ε, να δούμε το ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια εποχή όπου το γάλα de facto στο ράφι του σούπερ μάρκετ ε, είναι το φτηνότερο ποτό αναλύτρο έτσι, σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Και υπάρχουν λοιπόν πολλές προκλήσεις που πρέπει να α, λύσουμε. Και ξέρω πως πηγαίνω κόντρα στο ρεύμα, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε σε ποιο βαθμό θα πρέπει να κάνουμε καινούργιε σκέψεις για περισσότερη διασφάλιση κινδύνου, αλλά υπάρχουν και άλλα μέσα που είχαν αποδειχθεί πάρα πολύ καλά στο παρελθόν ή όταν μιλάμε για τα φυτικά προϊόντα υπάρχουν κάποια ευέλικτα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ε, παραδείγματος χάρη αν έχουμε πολύ καλή σοδιά και πέφτουν οι τιμές ε, θα μπορούσαμε αυτή τη σεζόν να παράγουμε περισσότερα βιοκαύσιμα. Και έτσι θα μειωθεί η παραγωγή και θα ανεβούν οι τιμές των τροφίμων, κάτι το οποίο νομίζω είναι σημαντικό για τους αγρότες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να απαντήσω στον κύριο Άγνιου, τον πολύ καλό μου φίλο. Ευχαριστώ τον κύριο Άγνιου που αναφέρθηκε στο ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο είμαστε ευτυχεί που η κυβέρνησή μα επέτρεψε πενταετή ε, απολογισμό όσον αφορά εξισορρόπηση της φορολόγησης. Είχαμε καλό διαμεσολαβητή που προδιετίας διορίστηκε και δημιουργήσε πολύ καλύτερη πειθαρχία στον τομέα για τους, από τους γεωργούς μέχρι τους λιανοπολιτές. Έγινε μια αναθεώρηση των εργασιών του φορέα αυτού και θέλουμε να ενισχυθούν οι εξουσίες του αλλά είχαμε καλά αποτελέσματα στον αφορά το διορισμό αυτού του διαμεσολαβητού, του συμπίν του τομέα. Να σας πω κύριε Άγνιου, ναι, υπάρχουν διάφοροι πάρα πολύ καλοί δημοσιογράφοι που ερευνούν το θέμα, αλλά αν δεν λειτουργήσει όλη, για να λειτουργήσει η αλυσίδα σωστά των τροφίμων, χρειάζεται διαφάνεια στις τιμές. Δεν πρέπει να βασιζόμαστε στους δημοσιογράφους. Και πρόκληση για όλους μας είναι πώς εμείς σαν Γεωργοί μπορούμε να πετύχουμε καλύτερο επιμερισμό της προστιθέμενης αξίας. Τα τελευταία δύο χρόνια το συζητούμε αυτό. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη θέση μας στην όλη αλυσίδα. Θα δημιουργήσουμε, πιστεύω, καλύτερες συνθήκες μέσω συνεργασίας. Και για να συνεργαστούμε και να δημιουργηθεί η απαιτούμενη εμπιστοσύνη, χρειαζόμαστε ε, επίκαιρα στοιχεία. Και πολλά στοιχεία διαθέσιμα είναι ξεπερασμένα. Πολλά έχουν, είναι δύο μηνών. Όσον αφορά την κρίση του γάλακτος τα τελευταία δύο χρόνια είδαμε ότι είχαμε τεράστια σκηνή στην αγορά του γαλακτοκομικού τομέα. Χρειαζόμαστε σωστά στοιχεία, επίκαιρα. Όχι όσον αφορά τις πρώτες ύλες, αλλά και τα παραγόμενα προϊόντα. Έτσι δημιουργείται εμπιστοσύνη. Και οι εκπρόσωποι των γεωργών έχουν την ίδια εξουσία όπως οι λενοπολιτές, οι μεταποιητές Δημιουργείται έτσι εμπιστοσύνη και υπάρχει κάτι επιμερισμό των κερδών. Το είδαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάποιοι γεωργοί μπορούν να συμμετάσχουν στι ομάδε και μορφώνουν τι τιμέ, μπορούν να αξιολογήσουν το κόστο τη παραγωγή, ασκήθηκαν πάνω του παρόμοιε πιέσει, όπω ασκήθηκαν και στου παραγωγού των γαλακτοκομικών ε, προϊόντων. Ναι, και στον τομέα το, της προθεσμιακής αγοράς ε, είχαμε καλέ εμπειρίε τα τελευταία δύο χρόνια. Αν Θέλουμε να κινηθούμε στην προθεσμιακή αγορά και για τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το ερυθρό κρέα, όπω είπε και ο Σπένινγκ, χρειαζόμαστε ρευστότητα. Πώ πετυχαίνουμε ρευστότητα στην αγορά, δημιουργώντα εμπιστοσύνη. Πώ δημιουργούμε εμπιστοσύνη μέσω επικαίρων στοιχείων, μέσω διαφάνειας. Και αυτά τα επίκαιρα στοιχεία απαιτούνται Αυτή θα πρέπει να είναι άμεση απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαφάνεια στην αγορά. Και μετά νομίζω ότι μπορούν να λυθούν τα άλλα προβλήματα όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων. Σας ευχαριστώ. Και ο κύριος Πένιγκς, ο καθηγητής. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την άκρο ενδιαφέρουσα εκδήλωση αυτή. Έμαθα πολλά σήμερα. Ένα σχόλιο βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Ένα από τα μέλη του Κοινοβουλίου αναφέρθηκε στη διαχείριση του κινδύνου και αν αποτελεί λύση για ανισορροπίες δυνάμεων. Πιστεύω ότι η διαχείριση του κινδύνου εν μέρη ίσως να παίζει ρόλο σε αυτό, αλλά δεν αντικαθιστά ε, και τις ε, ανισορροπίες δυνάμεων στην αλυσίδα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το σχόλιο λοιπόν για τη εξυχνίαση αυτού. Δεύτερον, ακροθυγώς αναφέρθηκα στο εξή ότι στην Ευρώπη έχουμε έξοχες δυνατότητες έρευνας και πολλές πληροφορίες για τη διαχείριση του κινδύνου και πώς να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά ούτω ώστε να έχουμε οικονομικά βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Η κυβέρνηση της ΕΠΑ, οι οργανώσεις των ΕΠΑ χρησιμοποιούν τα δικά μας αποτελέσματα και τις έρευνές μας για να το πετύχουν αυτό. Το μόνο στο οποίο προηγούνται είναι ότι όταν εξετάζουν τις πληροφορίες πολύ γρήγορα εφαρμόζουν τα σωστά μέτρα σε επίπεδο εκμετάλλευση. Ο Επίτροπος έλεγε ότι δεν είναι σίγουρος ότι με κατανοούσε. Με τα χαράς να πιω ένα καφεδάκι μαζί του για να το εξηγήσω το πώς λειτουργούν τα πράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ίσως ήταν ενδιαφέρον να εξετάσουμε αυτή τη διαδικασία. Να πώς διαδίδονται οι πληροφορίες και πώς τα ερευνητικά κέντρα μπορούν να έρχονται σε επαφή με τις εκμεταλλεύσεις, ούτως ώστε οι γεωργοί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να μπορούν πραγματικά να ανταγωνιστούν και σε υποϊσότιμες συνθήκες. Γι' αυτό πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές. Ευχαριστώ πολύ την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Σε ό,τι φορά. τον καφέ, βλέπετε πώς είμαστε για να κεράσετε καφέ σε Περάμε τώρα στην ανακεφαλαίωση, στις τελικές παρατηρήσεις. Ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας, ο κ. Γκίσεν, πρώτα. Τρία πράγματα θα ήθελα να αναφέρω. Μπορώ να απαντήσω σε όλα. Αλλά κοινή μας άποψη ήταν ε, βεβαίως πως είναι διαφορετικό πράγμα η αποτυχία αγοράς από τη διαχείριση του κινδύνου. Βεβαίως ε, ε, περνάνε και αυτές μέσα από τις αγορές. Ήταν σημαντική πράγματι η παρατήρησή σας και ήθελα να το ξεκαθαρίσω τώρα. Αν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο για τις αγορές και το εμπόριο. Κοιτάξτε, υπήρχαν πάρα πολλοί συμμετέχοντες στην αγορά, οι οποίοι είχαν τελείως διαφορετικές ε, ε, εμπειρίες και σχεδόν ε, όλοι όσοι συνεργάζονταν με μεγάλες αλυσίδες είχαν αρνητικές εμπειρίες. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως πως ε, πρέπει να έχουμε κάποια εικόνα η οποία θα είναι εχθρική. Τέλος για αυτό το οποίο είπατε για την πιστοποίηση είναι τεράστιο θέμα. Βεβαίως αντικατοπτρίζει ακριβώς το ότι θέλουν οι επιχειρήσεις να είναι απολύτως σίγουρες για την ποιότητα του προϊόντος. Αλλά βεβαίως αν μπορέσει έτσι ο αγρότης να ενισχύσει την δική του την ε, θέση, το προϊόν αυτό πληρώνεται και παραπάνω. Ε, πρόκειται λοιπόν ε, και για μια πτυχή που αφορά την, διαφα... την διασφάλιση της ποιότητας και της προέλευσης και έχει και πολλά ωφέλη. Να κάνω μια τελική παρατήρηση. αφορά και την συζήτηση για την μεταρρυθμισή του 2020. Για κάναμε κάποιες πρώτες ε, σκέψεις ε, για να δούμε ακριβώς σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να πάει και η επόμενη μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής. Ε. Αλλά βεβαίως αυτό δεν ήταν η δουλειά μας εμείς να κάνουμε τώρα οδικό χάρτη. Θέλαμε απλά να φέρουμε κάποια σημεία για να ξεκαθαρίσουμε ότι εάν θέλουμε μια πραγματική διαρθρωτική άλλαγη στον τομέα της κατεργασίας αλλά και της ίδιας της γεωργίας ε, θα πρέπει να υπάρξει μια διοχέτευση θα έλεγα και μια σωστή κατεύθυνση αυτής της ε, αλλαγής. Και το θέμα είναι πώς θα βρούμε τους νέους οι οποίοι θα στραφούν στην γεωργία αύριο και τι στόχους θα έχουν για να αγκαλιάσουν με ενθουσιασμό αυτό το επάγγελμα. Για να ανταποκριθούν και στις απαιτήσει της ε, κοινωνίας. Αυτά και σας ευχαριστώ. Θέλετε να δώσετε μήπως το λόγο σε κάποιο άλλος μέλος της ε, ομάδας εργασίας σας. Υπάρχει δυνατότητα. Τέθηκε μία ερώτηση για τις οικονομικές αξίες. Ε, στην Ουγγαρία έχουμε από τις αυστηρότερες ομοθεσίες για τις αθέμετες εμπορικές πρακτικές που εφαρμόζεται εδώ και 7 χρόνια. Βρισκόμαστε στην 8η χρονιά και έγινε η έρευνα πριν την εκπόνηση της νομοθεσίας και πριν από 2 χρόνια. Και όντως υπήρχε μια βελτίωση σε ό,τι αφορά την κατάσταση. Η... Ε, ε, μου μας είπαν και για τις περιόδους ε, πληρωμής ε, βελτιώθηκαν τα πράγματα για τους παραγωγούς και ήταν πολύ σημαντικό. Βέβαια δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα της αλυσίδας εφοδιασμού, θέματα διάρθρωσης, θέματα των ε, εμπορευμάτων, των αλυσίδων ε, διανομής με τις ιδιωτικές ετικέτες. Τέτοιου του θέματα δεν επιλύθηκαν, αλλά είναι χρήσιμο το εργαλείο παρόλα αυτά. Δεν είναι όμως πανάκια για όλα τα προβλήματα των γεωργών. Σας ευχαριστώ. Ε, κυρία Σιρακούζα από το γραφείο του Επιτρόπου πριν να ξαναδώσω το λόγο στον Επίτροπο Χόγκαν. Όχι, δεν χρειάζεται. Ο Επίτροπος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά τους. Θεωρώ ότι διαμορφώνεται μια πολιτική από την Επιτροπή ότι υποστηρίζει τις συστάσεις και την έκθεση δικής ομάδας. Κάτι που καθησυχάζει τους εμπειρογνώμονες. Διάφοροι ομιλητές όπως κ. Μακίνες, κ. Κώστιγκερ, ο κ. Ντόρφμαν και ο κ. Ντες και άλλοι αναφέρθηκαν στην εφαρμογή των συστάσεων. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίστηκε στο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2017. Δεν προϋπήρξε κάτι τέτοιο. Βλέπετε προφανώς ότι θέλω να δω τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η θέση των γεωργών θα πρέπει να έχουμε και υποστήριξη. Να λάβουμε υπόψη απόψη του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και των άλλων επιτροπών. Δεν θέλουμε να αγωνατίσουμε στα σε κάποιον. Θέλουμε να κερδίσουμε την υποστήριξή του για να εφαρμόσουμε κάποια πράγματα που προτείνει η έκθεση. Το ίδιο και αφορά και τη Γενική Διεύθυνση Γκρό, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα να πετύξουμε υποστήριξη τη βιωσιμότητα του Γεωργού από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντο. Του απασχολεί η βιωσιμότητα άλλων τομέων. Η DG Grow, η DG.com και εμείς θα πρέπει να συνεργαστούμε για να συμφωνήσουμε. Και εσείς μετά και το Συμβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσετε για την περαιτέρω πορεία, την νομοθετική, για να βελτιώσουμε τη θέση του Γιωργού στην παραγωγή τροφίμων και στη σχετική αλυσίδα. Η κυρία Μαγκίνες ρώτησε ποια είναι η άποψη της ειδική ομάδας για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ήταν εκτός από την εντολή τους. Θέλω να γνωστοποιήσουν οι 12 εμπειρογνώμονες τις απόψεις τους. Δεν θέλω να σχολιάζω απόψεις που δεν σχεδιάζονται με για τη σύνταξη τη εκθέσεω. Το Δεκέμβριο, στι 5 Δεκεμβρίου, εξέφρασα απόψει για την τοχή τη αγορά, άμεσε πληρωμέ, βιωσιμότητα ε, και ελπίζω αυτά τα σχόλια να σα ικανοποιούν. Ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια του 2017 θα είμαστε θέση να υποβάλουμε προτάσεις θα συνεργαστούμε με άλλε μονάδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μας στηρίξουν στις προτάσεις μας που θα πορεύσουν από τις συστάσεις. Ο κ. Ράγκ αναφέρθηκε στα παρατηρητήρια για τα απορροκεπευτικά. Μετά την επέκταση των παρατηρητηρίων για περισσότερες πληροφορίε για το τομέα του κρέατος θα εξετάσουμε και άλλους τομείς όπως τα απορροκυπευτικά. Δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα σε μελλοντικέ προτάσεις. διότι πρέπει να λάβω πρώτα τις απόψεις που ακούστηκαν σήμερα εδώ. Η κυρία Πύρη, ε, υπάρχει, ε, διατίθεται στη Γεωργία ε, το ταμείο αυτό για τους νέους, η Ολλανδική κυβέρνηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει, υπάρχουν πλατφόρμες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβάνονται και οι Γεωργοί, για να ληφθεί υπόψη, να χρησιμοποιηθεί αυτή η χρηματοδότηση και ελπίζω ότι όταν ληφθούν νομοθετικής φύσεως αποφάσεις επί του θέματος, ότι και οι Γεωργοί πάντα θα έχουν τελικό λόγο όσον αφορά ε, τις αποφάσεις περί παραγωγής και όχι λιανοπολιτής. Δεν θα πρέπει να απολέσουν τη θέση τους οι γεωργοί. Για τις έρευνες, για τις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ ε, δεν μπορώ να σχολιάσω εφόσον διενεργούνται οι έρευνες. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία των ερευνών πρώτα. Ο κ. Φλάναγκαλ ισότιμους όρους ανταγωνισμού και το κόστος χρηματοδοτήσεως. Αλλά είναι και η διαθεσιμότητα, όχι μόνο το κόστος. Θα ξέρετε από τη χώρα μας που ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε δύο ε, πυλώνες στο τραπεζικό τομέα που δεν συνεργάζονται ε, τέλεια όσον αφορά το είδος του χρήματος που διατίθεται και το κόστος του χρήματος που διατίθεται στους γεωργούς. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεως να προβλέψει ε, την ύπαρξη ανταγωνισμού για, μεταξύ των τραπεζών για να μειωθεί το κόστος χρηματοδοτήσεως. Μειώθηκε σε κάποια κάτι μέλη κατά 6% για βραχυπρόθεσμα δάνεια μέχρι 2,9% για πιο μακροπρόθεσμα δάνεια, αλλά δεν είναι όσο ικανοποιητικό θα θέλαμε ώστε οι νέοι γεωργοί ή εκείνοι που ξεκινούν στη γεωργία να μπορούν να έχουν ένα λογικό κόστος να αντιμετωπίσουν για το χρήμα και να μην αντιμετωπίζουν τα επιτόκια που ε, προβλέπονται τώρα. Η κυρία Αγγιλέρα αναφέρθηκε στο θεμητό ανταγωνισμό όσον αφορά τι συμφωνίε Αφρική-Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Συμφωνούμε, αυτό συμβαίνει και κυρίω όσον αφορά την Ισία. Υπήρξε μεγάλη ανησυχία και στην Ιταλία και την Ελλάδα και την Ισπανία για τι μεγάλε ποσότητε ελαιολάδου που προσωρινά θα εισαγάγαμε για τα δύο χρόνια. Βέβαια δεν πραγματοποιήθηκαν τα όσα εκφράστηκαμε των ανησυχιών, διότι δεν ήταν ανταγωνιστικό το τυνησιακό προϊόν. Αλλά βέβαια ευνοήθηκε τελικά η Ισπανία από την όλη διαδικασία. Τελικά μπήκε πολύ μικρή ποσότητα. Ισότιμες συνθήκες απαιτούνται για να ανταποκρίνονται στα υψηλές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτή ήταν η θέση που ακολούθησα σε όλες τις διαπραγματεύσεις εμπορικές στις οποίες συμμετείχα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφέρθηκε η θέση των νέων γεωργών, το είπα Στι 5 Δεκεμβρίου στην ομιλία μου. ένα από του πυλώνε βιωσιμότητα, αντοχή της και παραγωγή, αναπαραγωγή μάλλον, προβλέπω στου διάφορες οργανώσει των νέων γεωργών να μα δώσουν προτάσει το 2017 και το 2018 σχετικά με του νέου παραγωγού. Δεν έχω λάβει πολλέ προτάσει, αλλά περιμένω προτάσει, προσβλέπω σε αυτό. Για το Eurocommerce να πω ότι αν 20 κράτη-μέλη κινηθούν από μόνα τους, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να το σημειώσει πολιτικός στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο ότι σημειώνεται η ύπαρξη προβλήματος και ανταποκρινόμεθα σχετικά μέσω και στις ακροάσεις. Καλωσορίζω την υποστήριξη που σημειώθηκε σήμερα στο φασιστάσεις για διαφάνεια της αγοράς και για την καλύτερη διοργάνωση των γεωργών. Αν μας λέτε ότι τα στοιχεία σχετικά με την προστιθέμενη αξία τα θέλετε, προσβλέπουμε εν ευθέτω χρόνο να μας δώσετε τα σωστά στοιχεία. Έτσι όλοι θα ενημερωθούμε στα πλαίσια των μελλοντικών συζητήσεων για να καταλήξουμε ισορροπημένα αποτελέσματα για τις σχετικές δράσεις. Εν γέννη, Πρόεδρε, μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένο με το συνέστημα που δημιούργησε η έκθεση. Με όσα εκφράστηκαν σήμερα λόγω της εκθέσεως, μου δίνει την πεποίθηση να κινηθούμε το 2017 για να αποκατασταθεί η σωστή θέση του Γεωργού στην αλυσίδα τροφίμων. Σας ευχαριστώ. Και πριν ευχαριστήσω όλους τους ε, συμμετέχοντες, ήθελα να κάνω λίγα σχόλια. Μιλούμε για την τροφική αλυσίδα που έχει τρεις βασικούς παράγοντες, το, παράγοντες τον γεωργό, τον μεταποιητή και τον έμπορο. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε την ισορροπία μεταξύ των τριών αυτών παραγόντων της τροφικής αλυσίδας, ώστε να εξυπηρετηθούν και οι τρεις παράγοντες και αυτό θα επηρεάσει και το κόστος παραγωγής στο επίπεδο του γεωργού. Επίσης, ε, πολύ σημαντικός είναι ο διάλογος μεταξύ των κρίκων αυτής της τροφικής αλυσίδας και ε, γι' αυτό νόημα έχει να έχουμε ανοιχτό, διαφανή και ειλικρινή διάλογο και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ε, διαφόρων μερών και παραγόντων αυτής της τροφικής αλυσίδας. Επίσης, η προσπάθεια καταπολέμησης της κερδοσκοπίας, γιατί κερδοσκοπία υπάρχει, υπάρχει κερδοσκοπία στις αγορές. Και θα πρέπει πρώτα αυτό να χτυπήσουμε, τους κερδοσκόπους, ε, την κερδοσκοπία και μετά να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα στοιχεία της αλυσίδας της τροφικής. Επίσης, μιλήσαμε για τα προβλήματα που έχουν οι γεωργοί στη συνεργασία τους ε, ή στην οργάνωσή τους. Πώς θα εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση στις οργανώσεις, μεγαλύτερη συγκέντρωση της παραγωγής θα πρέπει να συνεργάζονται αυτοί οι επιμέρους οργανισμοί γιατί έτσι θα ενισχυθεί το βάρος τους, το ειδικό τους βάρος στην αγορά. Μιλήσαμε για την παγκόσμια αγορά, για την ευρωπαϊκή αγορά και γι' αυτό χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές λύσεις ή παγκόσμιες λύσεις. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό ότι οι λύσεις θα πρέπει να βρεθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό περιμένουν από εμά οι Γεωργοί. Φυσικά υπάρχει ε, το πρόβλημα πώς θα ε, υποβάλλουμε αυτές τις προτάσεις για ευρωπαϊκές λύσεις. Γιατί υπάρχουν και εξωτερικοί παράγοντες που μας επηρεάζουν και για να αντιμετωπίσουμε τους εξωτερικούς παράγοντες θα πρέπει να επιτύχουμε κάποια συμφωνία και σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί αυτοί οι εξωτερικοί, εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν τρομερά και την ανταγωνιστικότητα και τις ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου. Θα πρέπει λοιπόν να τις λάβουμε υπόψη. Επίσης, τα στοιχεία, τα δεδομένα αυτά που θα πρέπει να αποτελούν ε, ιδιοκτησία του δημοσίου, να είναι ε, δημόσιο αγαθό και να εξασφαλιστεί έτσι μεγαλύτερη διαφάνεια της αγοράς και πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Επίσης, ε, και ο χρηματοπιστωτικός τομέας δεν μπόρεσε να αυτορυθμιστεί. είναι ευκολότερες Παρ' όλα αυτά ήταν ευκολότερες οι ρυθμίσεις ε, ε, στο χρηματοπιστωτικό τομέα και παρόλα αυτά επειδή δεν υπήρξαν ε, τέτοιες ρυθμίσεις σε γενικότερο επίπεδο αλλά επαφεθήκαμε στην αυτορύθμιση είχαμε την κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στο γεωργικό τομέα. Έχουμε την αστάθεια των τιμών, την ανισορροπία μεταξύ των κρίκων της παραγωγής. Θα πρέπει να ληφθούν λοιπόν κάποιες γενικότερες λύσεις. Επίσης θέλουμε ισχυρότερο ανταγωνισμό αλλά θεμητό ανταγωνισμό. Γιατί σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε τεράστια επιρροή από τις πολυεθνικές εταιρείε που έχουν ε, τεράστια ισχύ. Οπότε, ε, τι, ποιο είναι το τελευταίο επιχείρημα που μας έμεινε, είναι η θέσπιση του δικαίου. Μόνο με τη θέσπιση νομοθετικών διατάξεων θα ενισχύσουμε κάπως τη δική μας θέση απέναντι σε αυτές τις πολυεθνικές. Νομίζω ότι έτσι με την δημόσια αυτή ακρόση Κάναμε μια γενική επισκόπηση των βασικών θεμάτων, όπως είναι η μεγάλη αστάθεια και οι διακοιμάσεις στις τιμές, όπως είπε η κυρία Ντελέ, τα προβλήματα της τροφικής αλυσίδας, το θέμα των αθέμητων εμπορικών πρακτικών, για το οποίο ήταν η συγκήτρια η κυρία Μαγκίνες. Και για όλα αυτά είχαμε και εμείς ήδη πολύ καλές προτάσεις, αλλά θα συνεχιστεί η συζήτηση για το μέλλον της κοινή ζωρικής πολιτικής. Αλλά με τη σημερινή ακρόαση συγκεντρώσαμε ακόμη περισσότερες γνώσεις και επιχειρήματα. Ευχαριστώ θερμότατα την ειδική ομάδα εργασίας, την Task Force για τις ζωρικές αγορές. Παρακαλώ διαβιβάστε τις ευχαριστίες μας στον ασθενή και απόντα σήμερα ε, διευθυντή, τον κύριο Φερμέγερ. Ευχηθείτε του και περαστικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, καλεσμένους μας εμπειρογνώμονες και όλους ε, όσοι έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Ε, είτε είναι πραγματικά δύσκολο αυτό το θέμα. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την παρουσία του. Και μάλιστα είχαμε και την πολυτέλεια του χρόνου σήμερα, οπότε είχα τη χαρά να μπορώ να σας δίνω το λόγο χωρίς να χρειάζεται μετά να σας περιορίσω στη διάρκεια της ομιλίας σας. Και πραγματικά αυτή ήταν σχετικά πρωτοφανή κατάσταση να έχουμε τέτοια πολυτέλεια χρόνου. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ και τους ε, διερμηνείς και να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει στις 27, 25 Ιανουαρίου, 9 με 12.30 και 3 με 6.30. Και ε, στις 26 Ιανουαρίου το πρωί. Αν δεν έχουμε τίποτα στα διάφορα, ευχαριστώ και την γραμματεία, γιατί πραγματικά δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να έχουμε επαρκή χρόνο για τη συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλό σας βράδυ.